Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Αρχίζουμε. Ε, ημερήσια διαταξή έχετε. Ετήσεις τροποποίησης δεν έχω. Ανακοινώσεις Προέδρου θα τα βρείτε στο Cont News. Η συνεδρίαση μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Οι γλώσσες αναφέρονται επίσης. Την προειδοποίηση για την απεργία την έχουμε ακούσει κατά επανάληψη και ελπίζουμε παρά τα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εργασία μας. Συστάσεις των συντονιστών επίσης μπορείτε να βρείτε στις 26 Ιουνίου διανεμήθηκαν σε όλα τα μέλη. Δεν έχω λάβει ενστάσεις. Sind wir beim dritten Tagesordnungspunkt Entlastung, der zweite Versuch mit dem Rat und dem Europäischen Rat. Οι διερμηνείς... Ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βρισκόμαστε στην 37η μέρα της ε, διαμαρτυρίας μας κατά της μονομερούς επιβολής άδικων συνδικών από τη δίκη του Κοινοβουλίου. Λυπούμαστε λοιπόν, που θα σας ενημερώσουμε ότι η διερμηνία θα ε, ολοκληρωθεί στην προγραμματισμένη ώρα της συνεδρίασης. Στη συνάντηση με το Συμβούλιο, εκτός από το πρόγευμα, υπήρξαν και οι εργασίες διότι εργαζόμεθα επί ενός μνημονίου συνεννόησης, το οποίο μνημόνιο συνεννόησης θα υποστεί και τροπολογήσεις εκ μέρους μας και τα έχουν τα μέλη και οι συντονιστές σήμερα. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν περισσότερο από ποτέ. Έχει αρχίσει κάποια κίνηση στη συζήτηση με το Συμβούλιο. Ίσως ο κύριος Βάλι μπορεί να συστήσει, αλλά για τελευταία φορά πια, την μη χορήγηση απαλλαγή στο Συμβούλιο. Έχει το λόγο ο συγητή μα κύριο Βάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για δεύτερη φορά φέτος μιλούμε για την απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Και πάλι σα τονίζω το Κοινοβούλιο μου η Πρόεδρος διακόπτη. Βάλτε τα ακουστικά σας. Άρα, βέβαια. Έλεγα ότι και πάλι σα τονίζω ότι όταν το Κοινοβούλιο το μόνο ερετό θεσμικό όργανο από του πολίτες εν τι τις προ προς το Συμβουλίο όσον αφορά τις δαπάνες είναι οι πολίτες ενδιαφέρομενοι οπότε γι' αυτό είναι σημαντικός αυτός ο διάλογος και γι' αυτό Θεωρούμε ότι είναι καθόδες το θέμα, άρα θα πρέπει να επιληθεί το συντομότερο. Παρ' όλα αυτά, το Συμβούλιο, όπως κάνει τις τελευταίες χρήσεις, δεν έχει ακόμη απαντήσει στις παρατηρήσεις μας. Ε, τι ψηφίζαμε το 18 Απριλίου. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των διοικητικών δαπανών και θα πρέπει αποτελεσματικά να γίνεται διαχείριση των χρημάτων των πολιτών. Και αυτό πρέπει να ισχύει για όλους. Σε αυτή τη δεύτερη έκθεση θέλω να τονίσω πρώτα-πρώτα αυτό το οποίο έχουμε γραμμή. Έχουμε ακόμα τις παρατηρήσεις τις σχετικές με το τι έχει γίνει με την διαμεσολάβηση όσον αφορά την διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας στο Συμβούλιο και το αίτημα να γίνει διαχωρισμός του προπολισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το Συμβούλιο που το έχει επαναλάβει στα, στις προηγούμενες το Κοινοβούλιο δεν έχει ληφθεί υπόψη. Έχουμε τώρα τις ε, διοργανικές συμφωνίες για να υπάρχει αυτό το Μητρό Διαφάνειας και όλα αυτά πάνε καλά και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο για τα ακίνητα παρά τις ανταλλαγές πληροφοριών των δύο θεσμικών οργάνων το Συμβούλιο συνεχίζει να μην παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με αυτά. Οπότε θα πρέπει να έχει προσβασιμότητα ο πολίτης στις σχετικές πληροφορίες και εμείς που τον εκπροσωπούμε. Άρα θα πρέπει να ενημερώσει το Συμβουλίο όσον αφορά την πρόοδο των πραγμάτων όσον αφορά τα ακίνητα και επίσης ε, κατά να αναφέρει τι γίνεται με τις δαπάνες. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, ιδίως όσον αφορά το ακίνητο, το κτίριο Ευρώπη. Στο δεύτερο κομμάτι του κειμένου έχω κάποιες επικρίσεις όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση και λέω ότι το Συμβούλιο θέλει να υπάρξει μια λύση όσον αφορά την απαλλαγή σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Οπότε πρέπει να υπάρχουν επικοδομητικές διμερείς ε, διαπραγματεύσεις και να υπάρξει αμοιβαία αποδεκτή λύση. Να είναι διακριτή η ρόλη των δύο θεσμικών οργάνων σε αυτή τη διαδικασία της απαλλαγής. Και σας υπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος επί των δεπάνων όπως τα άλλα θεσμικά όργανα και αυτό ήταν βάση της συμφωνίας του Ιανουαρίου του 2014 και είπαμε ότι έτσι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ε, επί τη βάση των παρατηρήσεών μας και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε για να υπάρχουν εγγυήσεις εύρυθμης λειτουργίας. Νομίζω ότι θα υπάρξει ε, περιθώριο για να συνεννοηθούμε και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση χρηστής διαχείρισης αλλά και διαφάνειας σε αυτή τη διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και βέβαια ό,τι διευκρινής θέλετε προθύμως θα σας παράσχω. Πρόεδρος. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Την έχετε την έκθεση προθεσμία καταθέσεων τροπολογιών 2 η ώρα της 10 η Σεπτεμβρίου. Σημειώνω ότι το Συμβούλιο εμένει στην αρχική του θέση. Δηλαδή ότι η συνθήκη προβλέπει απαλλαγή μόνο για τον προϋπολογισμό της Κομισιόν. Δεν είμαι βέβαιος εάν το θέμα του διαχωρισμού του προϋπολογισμού του Συμβουλίου από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο μπορεί να επιληθεί. Κατανοώ εξάλλου το επιχείρημα του Συμβουλίου, ότι δεν θέλει δηλαδή να ασκούμε πολιτική πίεση επί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσω της απαλλαγής του προϋπολογισμού. Διότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι και μία από τις ιερές αγελάδες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διότι δεν θέλουν να ασκείται πίεση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Το κατανοώ λοιπόν αυτό και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικές και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την απέτηση αυτή. Νομίζω ότι η τρέχουσα διαδικασία και η συνεννόηση με το Συμβούλιο, αν, ε, αν επιμείνουμε σε αυτό, μάλλον τίθεται σε κίνδυνο παρά να προχωρεί. Χρειάζεται βεβαίω περισσότερη διαφάνεια, σε αυτό συμφωνώ, αλλά επί του παρόντο θα είναι δυσχερέ. Α το πω έτσι. Να επιμείνουμε τόσο πολύ σε κάτι. Α, με συγχωρείτε, ο κύριο Αλαφράνκα είναι πρώτο και μετά ο κύριο Κλίντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βάλη για το έργο του στην έκθεσή του. Για αυτό το ιδιαίτερα πολύπλοκο και επίμαχο θέμα της απαλλαγής ε, του προπολογισμού του Συμβουλίου. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στη συζήτηση αυτή ότι το Κοινοβούλιο είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να κατανοήσουμε το ρόλο του Συμβουλίου ως οργάνου Νομίζω ότι το είπε και ο εισηγητής στην εκθεσή του ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ ε, των διάφορων αρμοδιοτήτων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου προκειμένου να υλοποιούν τις αρμοδιότητες δυνάμει των συνθηκών. Πάντοτε είχαμε δυσκολίες μεγάλες σε ό,τι αφορά την έγκριση αυτής της απαλλαγής και όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε σαφή έλλειψη συνεργασίας του Συμβουλίου. Και αυτό μας οδήγησε να αρνηθούμε την απαλλαγή 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2015. 14 και 15. Η διάσκεψη των Προέδρων δημιούργησε ένα μηχανισμό βάσει του οποίου αυτή η Επιτροπή πρέπει να κάνει επαφές με το Συμβούλιο για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι η έκθεση του κυρίου Βάλη επισημαίνει ότι υπάρχει μία σειρά σημαντικών εκρεμών ζητημάτων. Το Συμβούλιο συνεχίζει χωρίς να παρουσιάζει ξεχωριστό προπολογισμό μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνεχίζει να μην μας δίνει λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με την κτηριακή πολιτική στην ετήσια έκθεση και νομίζω ότι είναι καλή η πρόταση του εισηγητή ως προς την ε, διάκριση να έχουμε ε, λεπτομερείς ε, πληροφορίες για τους ανθρώπινους πόρους. Πιστεύω ότι στην έκθεση ικανοποιητικά αναφέρεται το θέμα των τρέχουσών διαπραγματεύσεων για να ενισχύσουμε το Μητρό Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούνιο είχαμε ένα διοργανικό διάλογο προκειμένου να ενισχύσουμε το Μητρό Διαφάνειας και πιστεύω ότι η έκθεση του κυρίου Βάλλη τοποθετείται στην παραδοσιακή γραμμή που ακολουθεί το Κοινοβουλίο μας. Όπως υπενθύμισε και η Πρόεδρος, ε, έχουμε μια προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Θα σκεφτούμε πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε την έκθεση αυτή η οποία μας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα λογική και συνεκτική και σέβεται πλήρως τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Θα δούμε πού θα καταλήξει και ο διοργανικός διάλογος, να δούμε αν το Συμβούλιο θέλει να κάνει κάποια προσπάθεια ως προς το να αναγνωρίσει τα προνόμια και τις αρμεδιότητες του Κοινοβουλίου σε σχέση με το θέμα της απαλλαγής, όμως σε κάθε περίπτωση, και για να κλείσω Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του, νομίζω ότι τοποθετείται σε μια γραμμή σεβασμού των προνομίων του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Κόν. Ο κύριος Κόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε που καθυστέρησα λίγα λεπτά να προσέλθω. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βάλη για την εργασία του που δεν είναι και απλή διότι και το θέμα δεν είναι απλό. Παρ' όλα αυτά άκουσα ότι από την χθεσινή συζήτηση προέκυψαν κάποια θετικά σημάδια, αν και όχι ακόμη λευκός καπνός. Θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στις διάφορες ε, σκέψεις που θα κάνουμε ότι υπάρχουν κάποιες θετικές τάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα συμφωνήσω με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά το ότι σήμερα δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να χορηγήσουμε απαλλαγή, διότι ελείπουν ακόμα σημαντικές πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, είναι επίσης σημαντικό τα θετικά αυτά σημεία τα οποία λάβαμε, τα θετικά μηνύματα τα οποία λάβαμε, να τα λάβουμε υπόψη, διότι μπορεί στο προσεχές μέλλον να αλλάξει η τοποθέτηση αυτή. Ο κ. Κλίντς. Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω πολλά στα σχόλια που μόλις ακούσαμε. Ο κύριος Βαλή έχει συντάξει μια ιδιαίτερα εξορροπημένη έκθεση που περιγράφει τα προβλήματα. Πρόκειται και για μια μακρά και ατυχή εξέλιξη. Είμαι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού ήδη από την αρχή του έτους. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκε επί μία δεκαετία να αρνούμεθα την χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο, διότι δεν δέχεται νόμιμα δικαιώματα εξουσίας του Κοινοβουλίου. Το ότι άρχισε χθε μια περίοδο ύφεση, α το πούμε έτσι, στη σχέση των δύο οργάνων, έχει καλώ. Αλλά μιλούμε για το 2016. Δεν μιλάμε καν για το 2018 ή 2017. Για το 2016 δεν είχε αλλάξει απολύτω τίποτε ακόμη. Ό,τι λοιπόν βελτίωση και αν υπάρξει, δεν θα πρέπει να οδηγήσει ώστε αναδρομικά να αλλάξουμε την κρίση μας. Το κακό, το άσχημο για μένα δεν είναι ότι υπάρχουν διαστάσεις απόψεων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ίσως σε κάποια επιμέρους θέματα να έχει διαφορετική άποψη το Συμβούλιο. Για μένα από τη συμπεριφορά του Συμβουλίου προκύπτει μια καταρχήν περιφρόνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δικαιωμάτων του. Και εγώ το βρίσκω αυτό πραγματικά λόγω συναγερμού για μας, διότι εμείς είμαστε εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης. Και τέτοιου είδους περιφρόνηση απέναντί μας είναι πραγματικά απαράδεκτη. Εάν διαγράφεται κάποια αλλαγή προς το καλύτερο, ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ. Είναι όμως και απολύτως αναγκαία η στάση αυτή αλλαγής, διότι ούτως αλλαγή, αντιμετωπίζει τόσες και τόσο μεγάλες προκλήσεις η Ευρώπη, που δεν μπορεί να αποδώσει εάν τα θεσμικά όργανα δεν λειτουργούν με σεβασμό τα μεν απέναντι στα δε. Για αυτό το λόγο λέω, καταρχήν έχει καλός, εάν επιτύχατε κυρία Πρόεδρε χθε να αρχίσετε να σπάτε λίγο τον πάγο, πολύ καλά. Όμως ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ώστε για το 2016 ξαναλέω να μπορούμε αναδρομικά να δώσουμε την απαλλαγή δεν μπορώ να αναλάβω τέτοια ευθύνη. Ελπίζω στο μέλλον να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά πρέπει να καταστήσουμε σαφέ απέναντι στο Συμβούλιο ότι τέτοιου είδου περιφρόνηση και έλλειψη σεβασμού δεν μπορούμε να δεχθούμε πλέον. Μην ανησυχείτε δώρα, δεν πρόκειται να κάνουμε, λέει η Πρόεδρο. Η κυρία Αιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο συνάδελφος Κον. και θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ανησυχία μου. Φυσικά ε, θα θέλαμε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα, αν όχι για φέτος αλλά τουλάχιστον για του χρόνου, να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ανάκτηση του διοργανικού παιχνιδιού με θετική έκβαση για τους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, με ανησυχεί επίσης ότι αυτές τις ημέρες γίναμε μάρτυρες μιας απαράδεκτης κατάστασης. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος ε, του Συμβουλίου ε, ουσιαστικά δεν ε, διευκολύνει τις συνεδρίες της. Συγγνώμη, μάλλον δεν υπακούει στην εντολή του για να διευκολύνει τη διακυβερνητικό παιχνίδι και αρνήθηκε να φιλοξενήσει ε, μία συνεδρίαση που είχαν ζητήσει μία σειρά κρατών μελών. Κοιτάξτε, δεν ε, είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν, αλλά στις ε, περιπτώσεις αυτής θα πρέπει να παρέμβουν. Δεν μπορεί να πει το Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Συμβουλίου ότι ε, μου ζητάνε 16 ε, κρατημέλη να συνεδριάσουν και να αρνείται. Θα πρέπει να δεχτεί το Συμβούλιο ότι η εντολή του είναι να διευκολύνει τις διοργανικές σχέσεις και μάλιστα τα καθήκοντα του Συμβουλίου. Δεν μπορεί δηλαδή να πει στα κρατη δεν θα συνεδριάσετε εδώ να πάτε απέναντι και δεν του κοστίζει τίποτα και μάλιστα είναι και υποχρέωσή του. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να του γίνει κάποια υπενθύμηση ότι εδώ δεν ε, πρόκειται ε, απλώς ε, για μια ευγενική ανταλλαγή σχέσεων, αλλά ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο ποιε είναι οι του. δεν μπορεί ας πούμε με αυτόν τον τρόπο ε, να απορρίπτει ένα αίτημα 16 κρατών μελών. Πρέπει να του υπενθυμίσουμε ότι δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα είναι σωστό η διαδικασία απαλλαγής να μην θεωρηθεί ως μοχλός. Βέβαια να λυθούν όλα τα προβλήματα νομίζω θέλει δύσκολο. Πάντως, κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί στη διαδικασία χωρίς απαλλαγή. Και εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Ο κύριος Βάλλη μπορεί να λάβει το λόγο, εκτός αν υπάρχει εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Ήθελα να ρωτήσω εν πάση περιπτώσει, αν και δεν το περίμενα να υπάρχει. Κύριε Βάλλη. Ευχαριστώ όλους τους ε, σκιώδους συζητητές. Πιστεύω ότι υπάρχει ξεκάθαρη σύγκληση, καθώς το θέμα το συζητάμε εδώ και χρόνια. Είμαστε όλοι αρκετά ικανοποιημένοι που φαίνεται να οδηγούμαστε σε κάποια λύση. Προφανώ θα πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε την πίεση, δηλαδή να ακολουθήσουμε την οδό που πρότεινε και η Πρόεδρος, αν θέλουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι ανησυχίες του κυρίου Κλίνς ε, είναι κάτι που συμμερίζομαι δηλαδή ότι μιλάμε τώρα για το 2016. Παρ' όλα αυτά, θα είμαι διαθέσιμος να συναντηθώ με όλους ε, τους εισηγητές. Αν ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα, ε, να μπορούσαμε να τα εντάξουμε στην έκθεση σε ένα ευρύ πνεύμα συμβιβασμού. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ερχόμαστε στο υπαριθμό 4, στον κύριο Τσέλερ αλλά δεν είναι ακόμη παρόν ο κύριος Τσέλερ, ο Εάν δεν έλθει αμέσω, θα πρέπει να συνεχίσουμε το υπαριθμό 5 και άρα τότε θα περιμένει. Όχι, few minutes δεν μου αρέσουν αυτά, λέει η πρόεδρος. Έρχομαι στο υπαριθμό 5. Τσερνόμπιλ, πυρηνική, ασφάλεια και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Καλώ ήρθατε κύριε Βιντ Νόβακ, διευθυντή του Τμήματος Πυρηνική Ασφάλειας τη ΕΤΑΑ. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Προέκυψε στην τελευταία συζήτηση στο σταθμό Ιγναλίνα, όπου στις συζητήσεις διαπιστώσαμε ότι έως τώρα ποτέ δεν έχουμε ασχοληθεί με το τι έγινε με τα ευρωπαϊκά χρήματα στο Τσέρνομπιλ και γύρω από το Τσέρνομπιλ και εάν θα πρέπει να προβλέψουμε καταβολές και για το μέλλον. Πληρωμές δηλαδή. Κύριε Νόβακ, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο για να μας πείτε περισσότερα για το Τσέρνομπιλ και από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, παρούσα είναι η κυρία Τόμελιν, η οποία διαχειρίζεται κονδύλια για την πυρηνική ενέργεια και θα χαρούμε πολύ αν μπορεί να μας διευκρινίσει τα σχετικά. Εσείς τώρα κύριε Νόβακ. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Thank you very much for your invitation. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας μιλήσω σε εσά την σημαντική σας επιτροπή. Η τράπεζα έχει ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση και τα γνωρίζετε και έχουμε τα τρία προγράμματα παύση λειτουργία σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία. Οπότε στην παρουσίασή μου που θα είναι σύντομη θέλω να εστιαστούμε σε κάποια άλλα έργα και προγράμματα που έχουμε χρηματοδοτήσει ως τράπεζα και όλα αυτά θα τα εντάξουμε ε, σε αυτό το ευρύτερο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην γειτνιάζουσα περιοχή. Επόμενη διαφάνεια. Δείξτε εδώ μία ματιά στο ιστορικό πλαίσιο. Όλα ξεκίνησαν με το ατύχημα στο Τσερνομπίλ το 1986. Πολλά χρόνια μετά από αυτό το ατύχημα η διεθνή κοινότητα προσπάθησε να βρει ε, πώς θα αντιδράσει από αυτή την πρόκληση, από ε, αυτούς τους κινδύνους που ενδημονούσαν ε, από αυτό το γεγονός. Και το ίδιο το Τσερνομπίλ ακόμα αποτελούσε πηγή κινδύνων. Οπότε το 1992 στη συνάντηση κορυφής του μονάχου των G7 ε, δημοσιοποιήθηκε ένα πρόγραμμα δράσης ώστε να βελτιωθεί η πυρηνική ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες ε, της πρώην Σοβιτικής Ένωσης. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε καινούργια μέσα πυρηνικής προστασίας σε συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις χώρες G7 και η τράπεζα συγκρότησε ένα επιτελείο ε, ούτως ώστε και από πλευρά τραπεζικής να καλύψουμε τα πράγματα και να κάτι σαν λογαριασμός και είχε ως προτεραιότητα το να υλοποιήσουμε το πώ θα εξυγχρονιζόντουσαν οι αντιδραστήρε σε διάφορε χώρε. το οποίο πρέπει να γίνει βράχη πρόθεσμα. Περιμέναμε δε ε, όλα αυτά να οδηγήσουν σε κλείσιμο τελικά αυτών των αντιδραστήρων. Οι, οι πολιτικοί ηγέτε τότε πιστεύουν ότι είναι θέμα λίγων ετών, όμω η εμπειρία κατέδειξε ότι τελικά χρειάστηκε πολύ μεγαλύτερη διαδρομή για να φτάσουμε εκεί. Θα προσπαθήσω τώρα να σας ε, ξεναγίσω σε αυτή την διατροπή, σε αυτό το μακρύ τελικά ταξίδι. Επόμενη διαφάνεια. Έχουμε τώρα 7 τέτοια ταμεία πυρηνικής ασφαλείας. Ε, πρόκειται για την ενίσχυση της υπόθεσης του κλεισίματος του αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ. Αυτός είναι ο βασικός ε, σκοπός, το πώς ο χώρος εκεί θα γίνει ασφαλής. Και βοήθησε πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Και πρόκειται για το πρόγραμμα NDEP, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο θα αντιμετώπιζε και θα ε, απέκλειε τους ε, κινδύνους όσον αφορά το περιβάλλον των ε, ε, κινήσεων των επιχειρήσεων του πυρηνικού στόλου της Σοβιετικής Ένωσης στην βορειοδυτική Ρωσία. Κάτι που είναι εξελίξη και επίσης μιλούμε για πρικοδότηση αυτών των 7 ταμείων που στα 5 δις ευρώ τα οποία εκταμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. η G7 και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πάμε στα 2,5 εκατομμύρια από τα οποία τα 2 δι, συγγνώμη, τα δύο δις αφορούν αυτά τα ταμεία και θα επανέλθουμε ε, ακριβώς με αυτών των κονδυλίων σε λίγο. Επόμενη διαφάνεια. δεν είναι τόσο ευκρινές, το συγγνώμη. Ε, εξηγεί το τι γίνεται με τις ε, ροές τις χρηματοδοτικές, τι γίνεται με όλα αυτά τα ταμεία, αυτά τα καταπιστεύματα και για να δούμε εδώ τώρα βασικά στοιχεία που είναι σημαντικά για την εργασία σας. Πρωταγωνιστικός ρόλος προβλέπεται για τους δωρητές, τα κράτη δωρητές με τα οποία κράτη συνεργαζόμαστε υπό όρους διαφάνειας. Και το τι γίνεται σε αυτά τα προγράμματα αποτελεί αντικείμενο λογοδοσίας προς τις ε, χώρες αυτές και όχι προς εμάς. Έχουμε χτές ε, διμερείς επαφές με αυτούς τους δωρητές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε εκπροσώπους της ε, εδώ και ιδίω για το Τσερνομπίλ έχουμε μια ad hoc ομάδα από την EBRD, από το, τις χώρες G7 και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελευταία επταετία έχουμε συνθεί πάνω από 50 φορές είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ το ότι όλα αυτά γίνονται με διαφάνεια και έχουμε αυτού του είδου την διαχείριση τη ε, χρηματοδότηση, για την οποία εμείς ε, εφαρμόζουμε κάποιο είδους ε, διαχείριση διαφύλαξης ακριβώς όπω διαχειριζόμαστε και τα δικά μας κονδύλια, τους δικούς μας πόρους. Οπότε τώρα έχουμε τόκους πάνω από 200 εκατομμύρια που έχουν επιστοθεί σε αυτά τα καταπιστέματα, σε αυτά τα ταμεία. Βέβαια λόγω των ισοτιμιών, λόγω των, ε, και της πολιτικής των αρνητικών επιτοκίων, όπως ε, ε, έχουν απομειωθεί αυτές οι εξοικονομήσεις αυτοί οι τόκοι. Πάντως δεν παίρνουν οι κυβερνήσεις των εμπλεκομένων χωρών επιπλέον χρήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό Και αυτό το λέω γιατί αποδεικνύει ότι υπάρχει έλεγχος των κοινωτικών πόρων. Τώρα, εξασφαλίσαμε ότι γίνεται αυστηρός έλεγχος και διαχείριση των τεχνικών διαδικασιών, των διαγωνισμών, προσφορών και αυτό είναι πιο δύσκολο από την διαχείριση των χρηματοοικονομικών γιατί χειριζόμαστε αυτά τα προγράμματα τα οποία για πρώτη φορά ε, τρέχουν και αυτά σε ένα θεσμικά δύσκολο περιβάλλον. Και ένα από τα αποτελέσματα που μας κάνει περήφανος, ιδιαίτερος περήφανος, είναι το ότι έχουμε συμβάσεις πάνω των 5 δις με αυτούς τους διαγωνισμούς. Και αυτά έγιναν ε, ξεκάθαρα και έντιμα. Επόμενη διαφάνεια. Για να δούμε τώρα σύντομα τι γίνεται με κάποια από αυτά τα προγράμματα. Να πάρετε μια γεύση της ουσίας του θέματος. Έχουμε αυτή την εταιρική σχέση της βόρειας διάστασης για το περιβάλλον. Ε, έχουμε αυτή, αυτό το κληροδότημα των επιχειρήσεων του Σοβιετικού Στόλου στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό που ήταν ε, κάτι το πάρα πολύ φρικτό και με αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να μειώσουμε τους κινδύνους, τους κινδύνους που εγκυμονούνται από αυτές τις τεράστιες ποσότητες ε, ε, ραδιενεργών αποβλήτων και πυρηνικών καυσίμων σε αυτό το τμήμα του Ατλαντικού. Οπότε και καταφέραμε να συμφωνήσουμε με τις Σοβιετικές Αρχές και έχουμε αυτό το στρατηγικό master plan του 2007 Οπότε έχουμε ε, πέραν άλλων μικροτέρων έχουμε τρία προγράμματα. Το Αντρέγεβα Μπέι που είναι μια εγκαταληφθήσα ε, ναυτική βάση. Ε, εκεί είχαμε δραστηριότητα για υποβρύχια. Το Λέψε επίσης ήταν ένα Και υπάρχει επίση ε, και άλλο πρόγραμμα που αφορά κάποιο υποβρύχιο ε, της Πάψα. Τώρα βλέπετε αυτή την εικόνα με τα πλοία, το Λάψα είναι αυτό το σκάφο το μεγάλο και έχει δύο ρημουλκά που το σέρνουν και ε, τότε που η φωτογραφία ήταν γεμάτο απόβλητα και καύσιμα βλαπτικά και ε, αυτό ήταν στο Μουρμάνσκ επί πολύ χρόνο. Θα σας πω τι έγινε τελικά. Στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε αυτό το οποίο ήταν το πιο ισχυρό πυρηνικό υποβρύχιο στον κόσμο. Ποιο ήταν το θέμα. Για άγνωστους λόγους αποσύρθηκε και το γεμίσανε με πυρηνικά καύσιμα. κυρίως από ουράνιο. Αλλά το πρόβλημα ήταν πώς θα αφαιρεθούν τα καύσιμα από το υποβρύχιο. Βλέπετε τώρα ένα άλλο σκάφος. Μεταφέρει τον Ιούνιο πέρσι κάποια καύσιμα από τον κόλπο Αντρέγεβα. Αυτό το πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα στη Ρωσία και συγκεκριμένα αυτό το πρόγραμμα για το κόλπο είναι ένα από τα παραδείγματα για το πώς αυτά τα καταπιστεύματα, αυτές, αυτές οι διμερείς εργασίε μπορούν να αποδώσουν πολύ καλύτερα από τις πολυμερείς προσπάθειες. την ε, Ιταλία, Νορβηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση του. Παρακάτω. Για να σας πω τώρα, ξεκινώντας από το Τσερνομπίλ. Μετά το ατύχημα, επί μία δεκαετία προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις για το πρόβλημα. Κρίσιμη καμπή απετέλεσε η πρώτη πολιτική απόφαση των G7 το 96. Αλλά μετά είχαμε το 97. Το Shelter Implementation ήταν ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε αυτές τις προσπάθειες και το 1997 μας ε, ζήτησαν οι χώρες G7 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκροτήσουμε αυτό τέλος πάντων το καταπίστευμα το CSF για το Τσερνομπίλ και άρχισε η εφαρμογή του, άρχισε η λειτουργία του 98. Να, η αφετηρία του προγράμματος. Βλέπετε πώς ε, ήταν ο αντιδραστήρας μετά το ατύχημα. Τι κληρονομήσαμε σε αυτές τις προσπαθίες μας 10 χρόνια αργότερα. Πάμε στο επόμενο. Βλέπετε εδώ τώρα ε, αυτό το, αυτή την κάλυψη, το shelter του 80, του 98, συγγνώμη, του 86, το 86. Εδώ έχουμε χιλιάδες τόνων που καλύπτει αυτός ο νάρθηγας. 20 τόνους από καύσιμα, πλουτόνιο. Σωστά φοβόταν ο κόσμος για το ότι θα μπορούσε αυτός ο νάρθηγας να καταρρεύσει και να έχουμε άλλη πυρηνική έκρηξη. Και μάρτυρες έχουν καταθέσει ότι το Politburo πίστευε ότι το 89 ακόμα ήταν δυνατόν να έχουμε το περίφημο φαινόμενο του συνδρόμου της ε, Κίνας. τέλος πάντων υπήρχαν μεγάλες ε, φόβος μεγάλων διαρών. Αυτά ήταν η αφετηρία μας. Για καταλάβετε κάπως το πρόγραμμα για αυτό το Νάρθηκα κάποιοι εμπειρογνώμονες με πόρους από την Ευρωπαϊκή Ζωή είχαν κάποιους στόχους ε, με την ασφάλεια, προγραμματικές αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν και θα έπρεπε επιστήμονες από πολλούς κλάδους να συνδυαστούν για αυτές τις αποφάσεις. αλλά τίποτα δεν έχει σχέση, τίποτα δεν, είχε προβλεφθεί ρητός για το θεσμικό περιβάλλον και την ε, υποδομή. Και είπαμε ότι το βεληνικές, το κόστος ε, θα καθοριζόταν μετά κάποια έρευνα και κάποιες προγραμματικές αποφάσεις. Γι' αυτό και έγινε κάποιο είδου αξιολόγηση αργότερα. Και ο αντιπρόσωπος της τράπεζας μου είπε τότε ότι αυτό είναι το πιο ρηψοκίνδυνο πρόγραμμα που υπάρχει. Πρώτη περίοδος. Σηματοδοτείται από αυτές τις προσπάθειες. Να προσθέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα και κατόπιν να βρούμε κάποιες λύσεις για τα πιο σημαντικά προβλήματα όσον αφορά ε, τη σταθεροποίηση του Νάρθη ή της σαρκοφάγου για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τα καύσιμα και αυτά τα υλικά που είχαν τα καύσιμα. Πολλά προβλήματα, πολλά τα εμπόδια για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Και διαφωνίες επίπεδο πολιτικών, μηχανικών. Ε, είχαμε και συγκρούσεις συμφερόντων εμπορικών, ε, βιομηχανίας, αλλά τελικά εξευρέθηκαν κάποιες ε, λύσεις που απέδωσαν. Το 2004 τελικά είχαμε τις συνθήκες για να αρχίσουμε να σταθεροποιήσουμε τις εγκαταστάσεις εκεί Και ο Πρωθυπουργό ενέκρινε το σχεδιασμό για αυτού του είδους την ε, προστασία της σαρκοφάγου. Να πως ε, εμφανίζεται τώρα η σαρκοφάγος μετά από τη σταθεροποίησή της και όλοι είναι ε, σχεδόν σίγουροι ότι έχει μειωθεί κατά 100 τουλάχιστον, 100 πλάσιο δηλαδή, η, ο κίνδυνος κατάρρευσης. Τώρα το επόμενο ήταν το New Safe Confinement νέα δηλαδή ασφαλής ε, οριοθέτηση του ε, αντιδραστήρα. Πέρασαμε τρία χρόνια μέχρι ότου γίνουν οι σχετικές ε, ε διαγωνισμοί και προμήθειες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημαντικά ορόσημα εν προκειμένου, όπως βλέπετε και στον πίνακα που δείχνω και οδηγούν στο, στην, στο, στην αποκορύφωση ας πούμε, που θα είναι τέλος του έτους του 2018, δηλαδή η παράδοση στο, στην Ουκρανία, στο κράτος της Ουκρανίας. Επόμενη διαφάνεια τώρα, το 2010-2011 εξακολουθούσαμε να αντιμετωπίζουμε την ε, βαριά ρήπανση στην περιοχή γύρω από τον αντιδραστήρα και η κατασκευή του τόξου έπρεπε να γίνει τουλάχιστον 250 μέτρα μακριά από τη σαρκοφάγο λόγω των επιπέδων ακτινοβολίας που είναι πάρα πολύ ψηλά πάνω από τη σαρκοφάγο. Ακόμα και εδώ λοιπόν οι εργολάβοι χρειάστηκε να απομακρύνουν τουλάχιστον 100.000 τόνους ε, χώματος και άμμου και να την αντικαταστήσουν με καθαρό υλικό. Άρχισε λοιπόν μετά η ε, κατασκευή, η συναρμολόγηση μάλλον της ε, αψίδας και το Σεπτέμβριο 2016 ολοκληρώθηκε η αψίδα 260 μέτρα στο βάθος και πάνω από 100 μέτρα ε, σε ύψος και αυτή μετακυλίστηκε πάνω από την σαρκοφάγο. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπει κανείς νωρίτερα φέτος ότι έχει τοποθετηθεί πλέον στην τελική της θέση, είναι λίγο πολύ έτοιμη η αψίδα πάντοτε και αναμένω ότι οι διάφορες δοκιμασίες που γίνονται θα ολοκληρωθούν μέχρι το Δεκέμβριο. Η δεύτερη κατάσταση τώρα στο Τσερνόμπιλ που συχνά σκιάζεται όμως από την άλλη είναι αυτή του αποπληρωμένου καυσίμου. Το αναλωμένο καυσίμου. Υψηλό ο κίνδυνο mm. εδώ, το ίδιο όπως ε, και η υψηλή ακτινοβολία της ίδιας της σαρκοφάγου, επομένω έργο κρίσιμο για την ασφάλεια, θα κοστίσει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ και στόχος μας είναι Ε, είναι δύσκολη η ιστορία και ο, αρχικός εργολάβος που είχε αναλάβει δεν μπόρεσε να βρει τις τεχνικές λύσεις. Χρειάστηκε λοιπόν να ξαναξεκινήσουμε το εγχείρημα από την αρχή. Η επόμενη διαφάνεια. Να λοιπόν η εικόνα που δίνει σήμερα η εγκατάσταση αυτή. Τώρα, εδώ βλέπετε τα σημεία, τους τόπους όπου θα τοποθετηθούν τα δοχεία διπλού ε, και τα οποία θα αποθηκευτούν εκεί για τα επόμενα 100 χρόνια. Έρχομαι τώρα στα χρήματα. Σύντομη εξήγηση για το πώς χρηματοδοτούνται τα προγράμματα αυτά. Το CSF, Shelter Implementation Plan, σε αριθμούς θα κοστίσει περίπου 2,100 δισεκατομμύρια ευρώ. Το New Safe Confinement είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Υπάρχουν και άλλα 250 συνολικά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται και ανέρχονται σε περίπου 600 εκατομμύρια και το κόστος. Το SIP, Shelter Implementation Plan, χρηματοδοτείται από το Ταμείο για το Τσενόμπιλ που είναι Ταμείο Δωρητών και το άλλο είναι ειδικό δάνειο της τράπεζας EBRD που έχει συνυπογράψει με το Ταμείο Τσερνόμπιλ και θα δείτε ότι η EBRD γίνεται ο μεγαλύτερος δωρητής για το Τσερνόμπιλ με καταβολή 750 εκατομμυρίων. Και τα χρήματα αυτά προέρχονται από το καθαρό εισόδημα της τράπεζας. Και το επόμενο, η επόμενη διαφάνεια, το ίδιο για την NSA. Έχουμε την εγκατάσταση του, των αναλωμένων καυσίμων που θα κοστίσει 215 περίπου εκατομμύρια και επίσης χρηματοδοτούνται από δάνειο της CBRD. Η επόμενη διαφάνεια εδώ δείχνω τη διαφάνεια αυτή την έφτιαξα ειδικά για την παρούσα συνεδρίαση, διότι νομίζω ότι δείχνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση και αντίθετα με, την, μεταδιεθνή τα διεθνή ταμεία για το decommissioning για την ε, πάυση δηλαδή λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων, έχουμε δώσει 98% του ποσού Εδώ ο προπολογισμό της Ένωση έχει συμβάλει κατά λιγότερο των 20% από το συνολικό ποσό. Ένα από τους ρόλους που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία είναι να ηγηθεί της προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων για το εγχείρημα αυτό. Όπως είπα, ήταν θετικό ο ρόλος της Κομισιόν και το αποτέλεσμα ήταν ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα ε, αποτέλεσαν αρχή για πάρα πολύ σημαντικό ποσό χρημάτων που προήλθαν από άλλες πηγές με μεγάλη γενοδορία από την τράπεζα EBRD αλλά και από άλλους δωρητές. Σημειώνω επίσης για τα αποκομιζόμενα επιτόκια συνολικά 170 εκατομμύρια και άλλα 100 εκατομμύρια από τόκους για το Decommissioning Fund. Υπάρχει και μια πρώτη τελευταία γραμμή για το συνολικό πόσο 45 εκατομμύρια που έλαβε το Ταμείο από τον εργολάβο ο οποίος δεν τα κατάφερε τελικά να βρει την τεχνική λύση για το έργο ISF και πήραμε πίσω τα χρήματα. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τα επιτεύγματα των ταμείων αυτών Δεν θα μιλήσω για το Διεθνές Ταμείο για την πάυση λειτουργία των σταθμών, αλλά λίγα για τα οικονομικά. Όταν κοιτάζω προς τα πίσω, από εκεί που ξεκινήσαμε, το 2001 με τα ταμεία αυτά. Κάθε άλλο παρά ορθές πρακτικές. Δεν είχαμε καμία από τις συνθήκες που ήταν αναγκαίες για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα decommissioning. Δεν σας τα πω όλα αυτά, αλλά δεν υπήρχε στρατηγική, δεν υπήρχαν σχέδια, δεν υπήρχε εθνική χρηματοδότηση, άλλη βέβαια κληρονομιά της Σοβιετικής ε, περίοδου, δεν υπήρχε τεχνογνωσία, ήταν, δεν υπήρχε ε, απογραφή των πυρηνικών σταθμών, επίσης τα ε, ρυθμιστικά πλαίσια ήταν απολύτως ανεπαρκή όλα αυτά κληρονομιά της Σοβιετικής περίοδου και υπήρχε και μια σημαντική υπόγεια αντίσταση στο κλείσιμο των αντιδραστήρων. Και αυτή συνεχίστηκε μέχρι που έκλεισε και ο τελευταίος αντιδραστήρας. Περάσαμε δύσκολες ιστορικά στιγμές. Όταν όμως βλέπω που βρισκόμαστε σήμερα, αισθάνομαι απόλυτα ικανοποιημένος. Έχουν κλείσει 8 8 υψηλού κινδύνου πυρηνικοί αντιδραστήρες όπως προβλεπόταν στα σχέδια. Η διάλυση των εγκαταστάσεων έχει προχωρήσει σε ένα σημείο που να σκεφτεί κανείς να τους ξαναβάλει μπροστά τους αντιδραστήρες αυτού δεν έχει κανένα νόημα πλέον. Έχει δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή, λίγα στοιχεία παραμένουν ακόμα σε φάση κατασκευής και με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας προφορώ ότι πέρασα από τη Βουλγαρία την προηγούμενη εβδομάδα όπου κατέστην Μάρτης της τελευταίας δοκιμασίας της εγκατάστασης για, το, για την τήξη του πλάσματος, το οποίο είχε πάρα, πέρασε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, όμως έχει δώσει πάρα πολύ καταπληκτικά αποτελέσματα με μεγάλο επίπεδο μείωσης στη διάρκεια της δοκιμασίας ο όγκος των ε, αποβλήτων μειώθηκε κατά 81 φορές. Πραγματικά τεράστια, πρωτοφανής επιτυχία για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων έχει αφαιρεθεί το καύσιμο από τους αντιδραστήρες. Άλλο ε, bullet point αυτό, όπως το είδε και η κυρία Γκρέσλε στην Ιγναλίνα. Ο αντιδραστήρας 2 αφαιρέθηκε το καύσιμο από αυτόν 15 μήνες πριν από την προβλεπόμενη χρονική στιγμή. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο διότι ήταν δύσκολη η μετάβαση αυτή και τώρα έχουμε πλέον οργανισμό για το decommissioning που είναι αποφασισμένοι, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τι κάνουν και αφοσιωμένοι στο σκοπό τους. Και ελέγχονται από πάρα πολύ ενισχυμένους πυρηνικούς ρυθμιστές πλέον στη χώρα αυτή. Παραμένουν βέβαια προκλήσεις, δεν έχει ακόμα τελειώσει η δουλειά μας μέχρι ότου να διαλυθούν τα κτίρια των αντιδραστήρων, μέχρι ότου αποθηκευτεί με ασφαλή τρόπο το ε, αναλωμένο καύσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η απειλή αυτών των αντιδραστήρων έχει απαλληφθεί για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Νομίζω όμως ότι είναι διαχειρίσιμο το έργο αυτό. Συνεχίζεται η συνεργασία. Η συνεργασία είναι καλή της Κομισιόν, της Ένωσης και των ε, χωρών ε, που είναι οι απολύτριες των κονδυλίων. Τώρα, πολύ σύντομα. Ε, έχουμε κάνει σημαντικές, σημαντικά βήματα πρόοδου. Έχουν μειωθεί κατά πολύ οι κίνδυνοι. Διαλύθηκε εκείνο το τεράστιο υποβρύχιο από τιτάνιο και έχει μετακινηθεί και το καψιμό του στο Μαγιάκ. Και το παγωθραυστικό Λέψε αφαιρούμε και εκεί το, ε, το πυρηνικό καύσιμο και μέσα στο 2018 θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή. Τώρα, η επόμενη διαφάνεια. του Τσερνόπιλ βρήκαμε λύσεις λοιπόν για τις προκλήσεις που προκύπτουν από το ατύχημα του Τσερνόπιλ και τις έχουμε εφαρμόσει. Θα είδατε ότι έχει σταθεροποιηθεί η σαρκοφάγος και το νέο κάλυμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αψίδα δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 2018. Το ίδιο η αφαίρεση του αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου και η επεξεργασία του στις νέες εγκαταστάσεις τις οποίες επίσης χρηματοδοτούμε. Και αρχίζει Σεπτέμβριο του 2018 η προσπάθεια αυτή. Στην επόμενη διαφάνεια. Α, δεν έχω άλλη. Έφτασα στο τέλος λοιπόν της παρουσίασής μου. Τώρα, σαν ας πούμε μια, ως μια καταληκτική παρατήρηση. Θα ήθελα να πω ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είτε άμεσα είτε ως συμβολή στο πολυμερές ταμείο μας είχαν τεράστια τεράστιες επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γειτονιά της σήμερα είναι πολύ ασφαλέστερος τόπος για να κατοικεί κανείς. σημαντικότατα πιο ασφαλής από ό,τι πριν από 30 χρόνια. Τουλάχιστον πυρηνικά, από πυρηνική πυρηνικές Τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιήθηκαν με αποτελεσματικό τρόπο. Στο ερώτημα αυτό η απάντησή μου είναι κατά κύριο λόγο ναι. Και έχω και τα στοιχεία για να την θεμελιώσω. Εν τέλει, Μπορούμε ωστόσο να είμαστε απόλυτα ήσυχοι σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια. Ασφαλώς όχι. Μία από τις βασικές αιτίες των ατυχημάτων που έχουμε υποστεί ως τώρα ήταν ο εφησυχασμός και η αγνόηση βασικών παραμέτρων της πυρηνικής ασφάλειας. Εκεί πρέπει να γίνει πολύ ακόμα εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νόβακ. Χαίρομαι που έχετε καλές ειδήσει. Πάρα πολύ εντυπωσιακή η παρουσίασή σας και απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πολύ θετικούς ρόλους. Και αυτός είναι από τους πιο συγκεκριμένους θετικούς ρόλους που έχω δει. Και σας συγχαίρω και προσωπικά είναι η τελευταία σας εμφάνιση σήμερα εδώ, το σημειώνω αυτό, διότι συνταξιοδοτήστε και γι' αυτό θελήσαμε να ε, έχουμε την ευκαιρία αυτή, να έχουμε κοντά μας τον ειδικό δηλαδή, ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει το τι έγινε τα τελευταία 25-30 χρόνια. Και βέβαια τις πολλές δράσεις που αναλάβατε. Νομίζω ότι μπορείτε να είστε ικανοποιημένος για τα όσα επιτύχατε. Θα ήθελα να δώσω τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο, στην κυρία Τόμαλιν, με την ερώτηση πέραν αυτών των χρηματοδοτήσεων που ανέπτυξε ο κύριος ε, Νόβακ, ποιες άλλες χρηματοδοτήσεις έχουμε σχετικά με πυρηνικά. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Εμείς δαπανούμε πολλά χρήματα στην Ουκρανία για παγκοσμίω για να ενδυναμώσουμε ε, την ε, πυρηνική νομοθεσία. Είναι αυτό κλειδί για τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, όπως είπε και ο κύριος Νόβακ, και για να αποφευχθούν τέτοια ατυχήματα να ξανασυμβούν στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τα απόβλητα, είμαστε ε, στην διαχείριση αποβλήτων, η δεύτερη ως προς τις δαπάνες και για το Τσερνόμπιλ. Στο Τσερνόμπιλ επίσης χρηματοδοτούμε κοινωνικά προγράμματα για να βοηθήσουμε τον ε, ντόπιο πληθυσμό να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του ατυχήματος, παραδείγματο χάρη. Έχουμε χρηματοδοτήσει έρευνα για την ε, θεραπεία του καρκίνου του θυροειδή, κυρίως στα παιδιά, και έχουμε ε, δημιουργήσει ε, ουσιαστικά ένα θερμοκήπιο για να παρέχουμε υγιή λαχανικά στον πληθυσμό και έχουμε φτιάξει και έναν αποτεφρωτή ξύλου έτσι ώστε να καίγεται με ασφάλεια ε, το μολυσμένο ξύλο, η μολυσμένη ξύλια. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έθεσε το ατύχημα και συνεχίζουμε να επενδύουμε παγκοσμίω στην πυρηνική ασφάλεια και ιδίω στο να ενδυναμώσουμε παγκοσμίω ε, την πυρηνική νομοθεσία και να ε, και επενδύουμε επίσης και στην διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Απάντησα στην ερώτησή σα. Κοιτάξτε, μπορείτε να μας δώσετε και αριθμητικά στοιχεία δηλαδή τα ποσά που έχουν επενδυθεί και τι θα επενδυθεί στο μέλλον σε αυτά τα project. Ίσως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε για να δούμε τι έχει δαπανηθεί στο παρελθόν και τι θα δαπανηθεί στο μέλλον. Σε σχέση με το τι έχει δαπανηθεί για το Ταμείο ε, για το εισαρκοφάγο, τα ανέφερε ε, περίπου 430 ε, ε, εκατομμύρια. Το νέο MFF ε, προβλέπει 300 εκατομμύρια ευρώ ως κονδύλι. Βέβαια αυτά δεν αφορούν την Ουκρανία μόνο, αλλά θα τα παρθεί Όποια χώρα δηλαδή ζητήσει βοήθεια στο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας ή των δικλείδων ασφαλείας, μπορεί να κάνει ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια θα υποφεληθεί από τη, βοήθειά μας στο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας. Στο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο λοιπόν έχουμε ένα νέο μέσο που θα λέγεται Ευρωπαϊκό Μέσο για την Πυρηνική Ασφάλεια, η INS, και ο προπολογισμό εκεί είναι 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει προτεθεί. Πρόεδρος, και κατόπιν έχουμε και την Ιγναλίνα που θα προσταθεί σε αυτό. Δηλαδή φτάνουμε στα 550 εκατομμύρια για περαιτέρω εργασίες για τους τρεις πυρηνικούς αντιδραστήριες. Αυτό έχει σχεδιαστεί. Η Ιγναλίνα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα γειτονίας. Πρόεδρος, ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί ε, χρησιμοποιείτε η DEFCO, μήπως μπορείτε να μας διαφωτίσετε για το θέμα αυτό ο μόνος ε, τόπος που ταιριάζει είναι εκεί. Δεν ε, ανήκει στη γαμαδέλτα ενέργειας. Υπάρχει ε, ουσιαστικά μια ιστορική ψημαχία για το που θα πρέπει να τοποθετηθεί, αλλά δεν ταιριάζει για τη γαμαδέλτα ενέργειας, γιατί δεν προωθούμε την πυρηνική ενέργεια, αλλά εδώ απλώς έχουμε θέμα πυρηνικής ασφάλειας και η γαμαδέλτα συνεργάζεται με τρίτες χώρες στο θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας και γι' αυτό έχει ενταχθεί στην ΤΕΦΚΟ. Επομένως, το ένα είναι θέμα της πρόθεσης και υπάρχουν και άλλα καθήκοντα που βλέπετε που ανήκουν αλλού, μάλιστα πολύ ενδιαφέρον. Εμπλώς ήμουν περίεργη για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, δεν έχει ζητήσει κανεί το λόγο. Α, συγγνώμη, κυρία Κάντερμπαχ, δεν είδα τον καταλογό μου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση ενός ε, ιδιαίτερα πολύπλοκου θέματος. Μας τα παρουσίασατε όλα με μεγάλη σαφήνεια. Από την άλλη, πραγματικά έχω εκπλαγεί που βλέπω πόσο λίγα γνωρίζουμε για όλα αυτά τα ζητήματα και η Επιτροπή Κόντ πραγματικά δεν ερευνά τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή της ενέργειας ε, είναι αντικείμενο διαχείρισης παγκοσμίω, αλλά αυτό το είδος παραγωγής ενέργειας, το είπατε και στο τέλος της παρουσίασής σας, ε, είναι κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να ελέγξουμε καθολικά. Επί της αρχής, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι τεράστιος και αν δούμε τα πραγματικά χρηματικά ποσά που πρέπει να δεπανηθούν ή θα πρέπει να τεθούν σε αποθεματικό για να μειώσουμε τους κινδύνους, αν αυτά είχαν επενδυθεί σε εναλλακτικέ μορφές ενέργειας, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα για την ασφάλεια των ανθρώπων και για την δημιουργία θέσεων εργασία. Έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια. Θα ήθελα να δω έναν αντίκτυπο στην επασχόληση, παραδείγματο χάρη. Γιατί αισθάνομαι ότι ε, έχουν αγοραστεί πάρα πολλά κρυβελικά, αλλά λίγα έχουν γίνει σε σχέση με τις θέσεις εργασίας. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει και με το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Θα ήθελα να δούμε και το θέμα της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας ε, λόγια, για την παρουσίασή μου, λέει ο κύριος Νόβακ. Θέσατε όμω ζητήματα που φυσικά είναι πολύ σημαντικά, αλλά ορισμένα υπερβαίνουν την εντολή μου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Οικοδόμησης και Ανάπτυξης είναι η μόνη πολυμερής ε, αναπτυξιακή τράπεζα ή μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει εντολή στο πυρηνικό τομέα, όμως αποκλειστικά στο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας. Έτσι λοιπόν, αν με ρωτήσουν ε, κάποιοι ποια είναι η θέση της τράπεζας, δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά των πυρηνικών, αλλά είμαστε υπέρ της πυρηνικής ασφάλειας. Και αν ε, είχαν διατηρηθεί οι προϋποθέσεις για την πυρηνική ασφάλεια, δεν θα είχαμε ούτε Τσερνόμπιλ ούτε Φουκουσίμα. Αυτό είναι το ένα. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της απασχόλησης, υπάρχουν ε, κάποιες επιπτώσεις, ανέφερα την εγκατάσταση περιπλάσματος. Αυτό βασίστηκε σε ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που δημιούργησε μια καινοτόμο τεχνολογία τουλάχιστον σε μισή ντουζίνα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα ασφαλής οριοθέτηση, New Safe Confinement στο Τσερνοβίλ, είναι μοναδικό τεχνολογικό και τεχνικό πρόγραμμα το οποίο για το οποίο συνεργάστηκαν επιστήμονες, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, πρόσωποι της βιομηχανίας από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ενώ θα μπορούσα να σας δώσω πολλά. Οι μεμβράνες που καλύπτουν τώρα την ασφαλή οριοθέτηση έπρεπε να σχεδιαστούν με έναν τρόπο ε, οι ταν διάφορες αντιφατικές απαιτήσει για την ανθεκτικότητα, την αντοχή, την ευελιξία και από ό,τι φαίνεται το υλικό που ήταν πιο κοντά σε αυτό ήταν το υλικό που χρησιμοποιεί ο γαλλικός στρατός για να σφραγίσει τις τορπίλες στα υποβρύχια. Όμως έπρεπε να αναβαθμιστούν τα υλικά. Επομένως, από τη σκοπιά της απασχόλησης, ακόμη και σήμερα, ο κύριος Ανάδοχος για τη νέα ασφαλή ροθέτηση απασχολεί πάνω από 2.000 ανθρώπους. Νομίζω ότι μπορεί να φέρει και τους 3.000. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νόβακ ε, για το έργο του και για τα τόσο θετικά αποτελέσματα που μας παρουσίασε σε ένα τόσο δύσκολο και πολύπλοκο ζήτημα. Φυσικά δεν μπορούμε να λέμε ότι αφενός χρηματοδοτούμε την πυρηνική ενέργεια και από την άλλη χρηματοδοτούμε την ασφάλεια για τη διαχείριση των αποβλήτων και σαν να ήταν μια αρνητική διαδικασία αυτή για τις ε, καρκινικές θεραπείες είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαχειριζόμαστε και να εργαζόμαστε με αυτή την ενέργεια. Επίσης έχουμε και το μεγάλο έργο να εργαζόμαστε στο θέμα της, ε, ενεργεια, της ενέργειας ε, σύνδεξης. Τώρα, ως προς την χρησιμοποίηση του προπολογισμού στην πυρηνική ασφάλεια, στον παροπλισμό και στην ε, παρακολούθηση του προβλήματος, γιατί το κύριο πρόβλημα είναι, παραδείγματος χάρη, η διαχείριση των αποβλήτων, όπως στην ενέργεια ε, των ορεικτών καυσίμων έχουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Κάθε ενέργεια έχει και αρνητικές πτυχές. το χάρη, τα αιωλικά πάρκα ε, έχουν ε, μια ένα αρνητικό οπτικό αντίκτυπο. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ξεκάθαρα ποια κονδύλια χρησιμοποιούνται και για ποιο λόγο ο κάθε προπολογισμό. Δηλαδή, να ξέρουμε σε κάθε τομέα για ποιο έργο και για ποιο συγκεκριμένο στοιχείο έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για να μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό και στους Ευρωπαίους πολίτες. Κύριος Μπαλτσίδης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με την ευκαιρία που μας δίδεται να ευχηθούμε καλή συνέχεια στον κύριο Νόβακ και είμαι σίγουρος ότι θα αξιοποιήσει τις ικανότητες του και κατά τη συνταξιοδότηση. Όντω υπάρχουν δυσκολίε όσον αφορά αυτέ τι ποινικέ εγκαταστάσει και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Από την αρχή που αντιμετωπίσαμε αυτά τα προβλήματα, ασχολήθηκε η Επιτροπή μας με αυτές τις προσπάθειες. Ακριβώς γιατί έπρεπε να ξέρουμε πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι. Έχω επισκεφθεί τρει-τέσσερι φορέ την πυρηνική εγκατάσταση εκεί και κατιαπίστωσα πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθούν τα σχετικά προγράμματα. Κατάλαβα γιατί κοστίζουν τόσο πολύ. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει ε, αφού καταμετρήσει πόσους πυρηνικούς συντηρητές έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπολογίσει το κόστος να δούμε πότε θα ε, κλείσουν ε, αυτές οι εγκαταστάσεις. Είχαμε θέσει ως όριο το 2020-2024, αλλά όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει πιθανότητα να μπορέσουμε να έχουμε καταφέρει οτιδήποτε τέτοιο πριν το 2040 και οι δαπάνες είναι πολλές. προωθείται η πυρηνική ενέργεια γιατί κοστίζει λίγο, θεωρείται καθαρή ενέργεια. Αλλά το, το θέμα δεν έχουν υπολογιστεί οι δαπάνε για τα πυρηνικά απόβλητα. Και το να έχουμε απόβλητα είναι κάτι το αναπόφευκτο. Οπότε, τι να σα πω, να μην με Πάντως πιστεύω ότι και στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την πυρηνική ενέργεια, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και να σκεφτούμε τις δαπάνες διαχείρισης των αποβλήτων. Να δούμε τι απαιτείται για κάθε πυρηνικό αντιδραστήρα και αυτά να τα αντιπαραβάλλουμε με το τι κέρδος έχουμε στην παραγωγή ενεργείας σε σχέση με άλλου τρόπου παραγωγής ενεργείας ή άλλου ενεργειακού πόρου τέλος πάντων. Κύριε Νόβακ, χωρίς μικρόφωνο, σας ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλέ ε, ε, απόψεις σε σχέση με αυτό που το οποίο είπατε. Υπήρξε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και η Επιτροπή σας όμως συνέχισε χωρίς να μείωσε τις προσπαθίες της. Ακριβώς όπως θα τα ξέρει και η κυρία Ρέστη μπορεί να σας το επιβεβαιώσει. Τώρα όσον αφορά το έργο της ε, τράπεζας. Πιστεύω ότι παρά την ε, ε, καθυστέρηση των προσπαθειών μας στην περίοδο 2009 έως το 2013 προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε σημείο όπου δεν θα είχαμε αύξηση των δαπανών. Πάντως είχαμε αυτή την ε, τετραετή καθυστέρηση. Άρα μείναμε στα πλαίσια των υπολογισμών μας ε, που είχαν γίνει πριν από 10 χρόνια. Είναι Λίνα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω του είδους του ποινικού αντιδραστήρα. Και ο αντιδραστής από γραφίτη είναι ιδιότυπος και απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Τελικά πάντως με ικανοποίηση βλέπω ότι ε, ε, ακολουθούνται αυτά τα οποία είχαμε πει και τα οποία πρέπει γίνει πολύ νωρίτερα. Και τελικά από κοινή προσπάθεια βρέθηκε μια κοινά αποδεικτή λύση. Αυτό είναι το μόνο ε, το οποίο ήταν σωστό να γίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, μια που έχουμε τέτοιους ε, αντιδραστήρες σε Ισπανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά θα πρέπει να τιμολογούνται ως ε, δαπάνες και στη φάση της ε, κατασκευής. Πρόεδρος. Πρέπει όντω να περιλαμβάνονται, να κοστολογούνται οι τιμέ αυτέ, εκτό αν έχει κανεί την ατυχία να κλείσει όπω η Ιγναλίνα νωρίτερα από ό,τι προβλέπετε. Σα παρακαλώ λοιπόν, σα ευχαριστώ πρώτον, σα εύχομαι καλή συνταξιοδότηση, με υγεία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και πάλι ε, σε κάποια ευκαιρία την αστήρευτη γνώση που έχετε για τα θέματα αυτά μια μακρά η συνεργασία μας. Έχουμε επισκεφτεί και τους τρεις αντιδραστήρες τους οποίους αναφέρατε. Εγώ προσωπικά σε κάθε περίπτωση που συναντηθήκαμε και συνεργαστήκαμε έχω εξέλθει με περισσότερη εμπειρία και γνώση. Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα και να μείνετε με διαβιές πνεύμα Τώρα κανονικά θα έπρεπε να ακολουθήσει ο κύριο Τσέλερ, διότι τελειώσαμε με το θέμα υπαριθμών 5 τη ημερησία διατάξεω. Πριν λίγο μόλι μου είπαν ότι έρχεται. Συνεχίζω τότε, λέει η πρόεδρο, με την ειδική έκθεση του υπαριθμών 6 δηλαδή, 8-2018 του ελεγκτικού συνεδρίου, για τις παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στην βιωσιμότητα. Η συγκεκριτή μας είναι ο κύριος Πυρίνσκι. Πρόκειται για σύντομη παρουσίαση της ειδική εκθέσεως. Είναι παρόν και ο αρμόδιος πάρεδρος του ελεκτικού συνεδρίου, κύριος Μπαλκό. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Από το 2000 στο 2013 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, είχε ε, προικοδοτήσει 75 δισεκατομμύρια ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις ε, σε επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, το να έχουμε βιώσιμα αποτελέσματα με τα χρήματα αυτά πριν από τα τέλη των project είναι σημαντικό για να, βοηθεί, για να έχουμε θετικά αποτελέσματα για του δικαιούχου και τις περιφέρειες. Αλλά σύμφωνα με μία μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα, την Επιτροπή σας το 2013, έχει υπάρξει μόνο περιορισμένο ενδιαφέρον από το δημόσιο τομέα σε ε, διαφορετικά ταμεία και ταμεία συνεχής ε, για το θέμα της βιωσιμότητας ε, και συνεπώς είναι διαθέσιμα μη πλήρη δεδομένα για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ εξετάσαμε στον ε, έλεγχό μας αν αυτά τα κονδύλια ήταν αντικείμενο διαχείρισης ε, με έναν τρόπο που να διασφαλίζει την ε, βιωσιμότητα των αποδάσεων και των αποτελεσμάτων και επίση εντοπίσαμε και του κύριου παράγοντε που αφορούν τη βιωσιμότητα. Για του σκοπού αυτού του ελέγχου, ορίζουμε τη βιωσιμότητα ω την ικανότητα ενό project να διατηρήσει τα ωφέλη του μακροπρόθεσμα όταν έχει ολοκληρωθεί το έργο και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την όμιμη περίοδο τη βιωσιμότητα. Τα ωφέλη ε, που ε, τα προγράμματα θα έπρεπε να παράγουν είναι ε, οικονομικά και χρηματοοικονομικά ωφέλη, επιστροφές ως προς το κόστος, αυξημένη παραγωγή, παραγωγικότητα, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καθώς και ε, περαιτέρω καινοτομία. Θα πρέπει επίσης να προσφέρουν μακροπρόθεσμα ωφέλη στις περιφέρειες όπου βρίσκονται η έννοια της βιωσιμότητας που χρησιμοποιήθηκε στον έλεγχο αυτό είναι επομένω ευρύτερη από την έννοια της νόμιμης βιωσιμότητας που έχει να κάνει με τις αποδόσεις ή με τα αγορασμένα περιουσιακά στοιχεία και καλύπτει μία μέγιστη περίοδο 5 ετών για τις μικρές και μικρές επιχειρήσεις όμως μόνο 3 έτη. Εξετάσαμε 41 πλήρη έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ μεταξύ του 2000 και του 2013 στην Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία. Στο πρώτο μέρος αυτού του ελέγχου αναλύσαμε την βιωσιμότητα των αποδόσεων και στο δεύτερο τμήμα τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που μπορεί να είναι έμεσα και άμεσα. Έμεσα και άμεσα και για τις αποδόσεις και για τα αποτελέσματα. Αξιολογήσαμε τη βιωσιμότητα στο τέλος ε, της ε, πενταετούς ή της τριετούς ε, περίοδου βιωσιμότητας και τη στιγμή του ελέγχου. Στο τρίτο τμήμα εντοπίσαμε τους κύριους λόγους γιατί οι παραγωγικές επενδύσεις πάσχουν σε βιωσιμότητα καθώς και σε, και σε πρακτικές. Βρήκαμε ότι μία πλειοψηφία ε, των σχεδίων είχε βιώσιμα αποτελέσματα. Ε, όταν είχαμε μερικώς βιώσιμα αποτελέσματα, αυτό οφειλόταν σε έλλειψη έμφασης ε, στην διαχείριση του υποστήριξη του ΕΤΒΑ σε παραγωγικές επενδύσεις μεταξύ του 2000 και του 2013 τα ε, project που ελέξαμε ε, γενικά είχαν αποδόσεις όπως είχε συνδυαστεί μόνο σε μία περίπτωση. Ε, ένας μηχανισμός δεν λειτουργούσε στο τέλος της νόμιμης περίοδου της βιωσιμότητας λόγω χρεοκοπίας. Στις περιπτώσεις περιπτώσεις, 31 περιπτώσεις, οι αποδόσεις υπήρχαν και λειτουργούσαν και τη στιγμή του ελέγχου. Σε 9 περιπτώσεις, δεν είχαν, ε, είτε δεν είχαν χρησιμοποιηθεί καθόλου, είχαν χρησιμοποιηθεί μερικώς, είχαν εγκατασταθεί από άλλο ε, από άλλο εξοπλισμό στο τέλος ε, της περίοδου αυτή η στάση μπορεί να αιτιολογείται από διάφορους λόγους πρέπει χάρη επειδή έπρεπε να αντικατασταθούν τα μηχανήματα ή συστήματα πληροφορικής λόγω φθοράς ή βλάβης για να αποκτηθεί πιο σύγχρονος εξοπλισμός ή λόγω αλλαγών στην ενεργειακή νομοθεσία οι απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νόμιμη βιωσιμότητα ε, ουσιαστικά πληρούνταν σε όλες τις περιοχές όπου υλοποιήσαμε τον έλεγχο. Στο τέλος της ε, περίοδου, πάνω από το ίμιση των project ε, εξακολουθούσαν να παράγουν αποτελέσματα πλήρως ή μερικώς. Όμως, για το υπόλοιπο ίμιση των έργων δεν μπορούσαμε να εξελογήσουμε πλήρως τη βιωσιμότητα γιατί οι πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες είτε δεν είχαν συλλεχθεί ή είχε λήξει η περίοδος αρχιοθέτησης. Τη στιγμή του ελέγχου τα περισσότερα έργα εξακολουθούν να παράγουν άμεσα αποτελέσματα όπως δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αυξημένη παραγωγικότητα. Όμως σε 8 ή ένα πέμπτο των 41 project που ελέγξαμε τέτοια αποτελέσματα δεν ήταν βιώσιμα και ήταν μόνο μερικώς βιώσιμο σε ένα, στο τέταρτο, δηλαδή σε 11 project ε, ε, συνολικά. Ε, από τις 19 υποθέσεις σε τρεις υπήρχαν κάποιοι λόγοι που δικαιολογούσαν την έλλειψη της βιωσιμότητας όπως το χάρη, εξελίξη στην αγορά, αλλά και στην εθνική νομοθεσία αλλά σε άλλες 5 περιπτώσεις η έλλειψη βιωσιμότητας οφειλόταν σε δυναμία στις διοίκηση, σε διαχείριση, σε άλλα προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις ίδιες τις ε, εταιρείε δικαιούχου. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι υπήρχαν κάποια δευτερογενή ωφέλη των project που είχαμε καλή βιωσιμότητα. Παραδείγματο ε, χάρη βοήθησαν τους δικαιούχους ε, να προβούν σε αναδιάρθρωση, να εξυγχρονίσουν ε, τα παραγωγικά περιουσιακά του στοιχεία, να προσαρμόσουν και να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια του προϊόντο να βελτιώσουν, ενισχύσουν την παραγωγικότητά του και τη θέση του στην αγορά αλλά να βελτιώσουν και την εικόνα τους και να υπάρχει καλύτερη πιστότητα από τους καταναλωτές. Επίσης, ωφελήθηκαν ε, από βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δάνεια και μπορούσαν να κάνουν περαιτέρω επενδύσεις με δικούς τους πόρους. Επίσης, ε, βρήκαμε κάποια έμεσα αποτελέσματα, ε, όπως περίπτωση χάρη αυξημένη απασχόληση, επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, περιβαλλοντικά ωφέλη, καινοτομία, αυτά δεν ε, είχαν ε, θεωρηθεί ως ρητή στόχοι για κάποιο από τα επιχειρησιακά προγράμματα ή τα project. Παρ' όλα αυτά, μια σειρά έργων συνεισέφερε σε τέτοια έμεσα αποτελέσματα. Ε, τα προγράμματα των οποίων τα άμεσα αποτελέσματα θεωρήθηκαν βιώσιμα Επίσης, είχαν κάποιες οικονομικές ή κοινωνικές θετικές συνέπειες για τις περιοχές ή τις τοπικές κοινότητες δημιούργησαν ε, μόνιμες ε, θέσεις εργασίας, είχαν ε, μεγαλύτερη στη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και σε υψηλότερους φόρους, αλλά υπάρχει και χαμηλότερη ρήπανση, ε, ήχορύπανση και απόβλητα η έλλειψη βιωσιμότητας μπορεί να οφειλόταν σε αλλαγές στην νομοθεσία ή σε την οικονομική κρίση, σε άλλες περιπτώσεις σε αδυναμίες της διαχείρισης. Αλλά ο κύριος λόγος ήταν ότι υπήρχε ανεπαρκής εστίαση στη βιωσιμότητα σε διάφορα επίπεδα διαχείρισης των κονδυλίων του ΕΤΠΑ. Τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν προωθούσαν αποτελεσματικά τη βιωσιμότητα και οι διαδικασίες επιλογής δεν λάμβαναν επαρκή υπόψη των συνθήκων για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Επίσης, ε, είδαμε ότι η απώλεια αποτελεσματικότητα δεν είχε ληφθεί υπόψη επαρκώς στην επιλογή των σχεδίων, γιατί οι διαχειριστικέ αρχές δεν θεώρησαν επαρκώς την ικανότητα των δικαιούχων να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι τα project ή να έχουν μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση μία ένδειξη τη απόλυτη αποτελεσματικότητα είναι όταν ένα ξεκινήσει πριν να δοθεί η επιχορήγηση και αυτό ήταν η περίπτωση σε έξι σχέδια. Σε τέτοιε περιπτώσει υπάρχει ο κίνδυνο οι δικαιούχοι που ε, οι δικαιούχοι θα είχαν ε, μπορέσει να υλοποιήσει τα προγράμματα χωρί ε, την επιδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρήκαμε μάλιστα και μία περίπτωση στην οποία ο δικαιούχος δήλωσε στην δήλωσή του ότι δεν θα χρειαζόταν ε, δάνειο ή επιχορήγηση για να εφαρμόσει το έργο. Και τέλος ε, βρήκαμε ότι 8 από τα αξιολογημένα προγράμματα θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί σε μια παρόμοια κλίμακα μόνο με ίδια κονδύλια των δικαιούχων ή αν έπαιρναν εμπορικά δάνεια χωρί να χρειάζονται και ευρωπαϊκέ επιχορηγήσει. Θεωρώ επομένω ότι η αν επαιρναν εμπορικα δανεια χωρίς να χρειαζονται και ευρωπαϊκές επιχορηγησει θεωρω επομενω είναι το αντίθετο τη βιωσιμότητα. Όχι μόνο δεν υπάρχουν καλά βιώσιμα αποτελέσματα που να χάνονται με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα αποτέλεσμα, γιατί τον λόγο αποτέλεσμα ε, θα είχε συμβεί ούτως ή άλλως. Και τέλος βρήκαμε ότι η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ε, ε, μετά το τέλος των project που δεν ήταν νομική απέτηση ουσιαστικά δεν υπήρχε ε, και δεν ε, εφαρμόστηκαν με συνέπεια τα διορθωτικά μέτρα αν και βελτιώθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ε, προγραμματική περίοδο 2014-2020, χρειάζεται περαιτέρω δράση για να πετύχουμε την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων. Και για την ε, περίοδο μετά το 2020, ο σχεδιασμό των προγραμμάτων ε, με σεβασμό στη βιωσιμότητα θα πρέπει να βελτιωθεί. Συστήνουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη καταρχήν να προωθήσουν βιώσιμα αποτελέσματα κατά το σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων, εστιαζόμενα περισσότερο στο να εντοπίσουν και να μετριάσουν του κινδύνου και ε, να ε, αναλύσουν περισσότερο τις ανάγκες, όπως την ανάγκη για δημόσια χρηματοδότηση, να βελτιώσουν ε, την διαδικασία επιλογής και τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο της απολύτως αποτελεσματικότητας, τρίτον, να δώσουν έμφαση στη βιωσιμότητα, στην παρακολουθήση και υποβολή εκτέσεων και τέλος, να καταστήσουν, να θεσπίσουν συγγνώμη ξεκάθαρα διορθωτικά μέτρα που σχετίζονται με την επιτεύξη των στόχων σε επίπεδο project δεκτό που υπάρχουν τέτοιοι στόχοι και να τα εφαρμόσουν συνεπώς. Επίση, συστήνουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερη προσοχή στο πώ τα κράτη-μέλη ε, αντιμετωπίζουν ε, τι ε, αποδόσει τη βιωσιμότητα και να διασφαλίσουν ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν σαφή διορθωτικά μέτρα σε ό,τι αφορά και τις διευθετήσεις ανάκτησης όταν τα project δεν σέβονται τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιβιωσιμότητας. Τέλος, η Κομισιόν μαζί με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις εξπόστε στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διερευνούν πιο συστηματικά τις διάφορες πτυχές ε, της βιωσιμότητας ε, των αποτελεσμάτων των project. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω εσάς κύριε Σεγητά και εσάς κυρία Πρόεδρε για την ενθουσιώδη στάση σας απέναντι στην έκθεση αυτή. Επίσης και εσάς κύριε Σεγητά για το πολύ ξεκάθαρο έγγραφο εργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Βρισκόμαστε λοιπόν την καρδιά των ε, προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομική ανάκαμψη. Ο κύριος Πυρίνσκι έχει το, λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στηρίζω απολύτως την άποψη που εκφράσατε. Πράγματι βρισκόμαστε στον πυρήνα των προσπαθειών και ιδίως του ελέγχου του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος της χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ευχαριστώ τον κύριο Μπάλκο, του συναδέλφου του, για την έκθεση που συνέταξαν και που ακόμη και από αυτή τη σύντομη παρουσίαση στην οποία προέβη φαίνεται καθαρά η πολύ σοβαρή δουλειά που έχει γίνει στην έκθεση αυτή σε βάθος έρευνες και χρήσιμες αναλύσεις και συμπεράσματα. Ε, από δύο φόρο τιμή στην εργασία αυτή τώρα για τις παραγωγικές επενδύσεις. Όλοι θα πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτή την έννοια των παραγωγικών επενδύσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που έχουν δαπανηθεί τα τελευταία, στην τελευταία προγραμματική περίοδο και να αναγνωρίσουμε ακριβώς τον ρόλο τον ρόλο κλειδί για όλους τους στόχους ανάπτυξη, βιώσιμη απασχόληση, μείωση ανισοτήτων που πρέπει ε, να είναι ο πυρήνας αυτών των παραγωγικών επενδύσεων. η ε, θεμελιώδεις στόχοι για να επιτευχθεί και η σύγκληση αλλά και η περιφερειακή και εδαφική συνοχή. Εν προκειμένου, ανησυχητικό είναι ότι στη διάρκεια των ελέγχων, σε ένα αριθμό υποθέσεων, δεν μπόρεσαν οι αρχές που διεξάγουν αυτές τις ε, επενδύσεις δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την αξία, την παραγωγική αξία των επενδύσεων. Ακούσαμε και τις ελλείψεις, ξεκινώντας από τον προγραμματισμό και φτάνοντας στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων και έτσι νομίζω ότι είναι σημαντικό να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις του κανονισμού κοινών διατάξεων και αυτόν που αρχίζει τώρα να ισχύει, αλλά και αυτόν που συντάσσεται. που θεωρώ ότι δεν περιλαμβάνουν διατυπώσεις που να πετούν, ας πούμε, κριτήρια ουσιοδών ορισμών της απόδοσης και των αποτελεσμάτων. Γιατί μόνο η επικέντρωση στην απόδοση, αν δηλαδή τα χρήματα τοποθετήθηκαν σωστά, δεν μας επιτρέπει να εξετάσουμε αν έχουν προκύψει και μακροπρόθεσμα βιώσιμα αποτελέσματα από τις επενδύσεις αυτές. Νομίζω ότι εδώ οφείλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, διότι δεν έλαβε υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2020-2027. Και ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη Περιφερειακής ανάπτυξη, εκεί χρειάζεται να υπάρχουν και δείκτε για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Μοιραζόμαστε τι ανησυχίε του ελεγκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά την διασφάλιση τη ικανότητα ιδίω μικρών και μεσών επιχειρήσεων, έχοντα υπόψη βεβαίω όλε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν και ιδίω όμω ό,τι αφορά την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους. Πρέπει να σκεφτεί κανείς τρόπους εξασφάλισης της βιωσιμότητας των μικρομεσών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις αρνητικές και θετικές εμπειρίες ε, της προηγούμενης περίοδου. Δεν αρκεί όμως αυτό, ε, διότι εν τέλει Οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε μια συνολικότερη βιομηχανική στρατηγική στο ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μεταφέρεται στα εθνικά επίπεδα με συμφωνίες συνεργασίας διότι μόνο τότε, εάν δηλαδή οι παραγωγικές επενδύσεις συναποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας μακροβιομηχανική στρατηγική μπορούν να παίξουν τον σωστό ρόλο. Τέλος, νομίζω κυρία Πρόεδρε, ότι υπάρχει λόγος να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τι χώρε μέλη να δεσμευτούν σε ένα εγχείρημα που θα σημαίνει ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν από την αρχή του σχεδιασμού του προγράμματος μέχρι την εκτέλεση των δαπανών, ώστε να παίξουν τον ρόλο που τους αρμόζει. Θα συμφωνήσω με το συμπέρασμα του κ. Μπάρκο ότι ο χρόνος που δαπανούμε εδώ στην παρούσα Επιτροπή για την εξέταση του θέματος αυτού είναι απολύτως δικαιολογημένος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νοβακόφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον σκιώδη εισηγητή του Λαϊκού Κόμματος, κ. Σταχόφσκι. Ευχαριστώ τον κύριο Μπάλκο πρώτα για την εργασία του, για την σύνταξη της εκθέσεως, καθώς και τον κύριο Πυρίνσκι για τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει για να μας υποβάλει έγγραφο εργασίας. Αυτά ξεπερνούν και το τα προγράμματα ERDF. Η βιωσιμότητα πρέπει να διατρέχει οριζόντια όλες οι ταπάνες του Ευρωπαϊκού προϋπολισμού και είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατευθύνει τις χώρες μέλη στην υιοθέτηση υψηλών προδιαγραφών για την εξασφάλιση βιωσιμότητας και προστιθέμενης αξίας της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βλέπουμε κατ' επανάληψη αδυναμίες διαχειρίσεως έργων που τελικώ οδηγούν σε σφαλμένη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τονίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει πιο συστημική προσέγγιση για την βιωσιμότητα των έργων. Χαίρομαι για τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου δεν αρκούν κατευθυντήρες γραμμές. Χρειάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων Σωστά είπε ο εισηγητή στο έγγραφο εργασία του ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει να εκτελούνται σωστά οι απαιτήσει, διότι καμιά φορά καταλήγουν αλλού τα χρήματα που προορίζονται τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται όπου αυτό είναι αναγκαίο. Δεν έχω άλλου που να ζητούν το λόγο, λέει η πρόεδρο, η κυρία Βάγνερ τη ε, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξη τη Επιτροπή. Ορίστε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και ευχαριστούμε για την παρουσίαση των κυρίων Μπάλκο αλλά και τον εισηγητή που μας τα είπε εξαντλητικά. Για να σταθούμε σε κάποια σημεία. Θεωρούμε πάρα πολύ θετική αυτή την έκθεση. Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι έτσι είναι πιο αποτελεσματική η έλεγχη σε σχέση με τα αποσπόμενα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική και όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων να έχουμε μέθοδο που να βασίζεται στα αποτελέσματα. Θέλουμε να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη βιωσιμότητα των ε, επενδύσεων για αυτή την περίοδο, σχέση με τις προηγούμενες συμφωνεί η Κομισιόν ότι πρέπει στο νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2020 να παρέχουν αυτές οι αρχές και τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται μια προσέγγιση στρατηγική όπως προβλέπει το πλαίσιο το 2020 είναι ξεκάθαρα αυτή η λογική παρέμβασης και έχουμε ε, προβλέψει διάφορα μέτρα μεταξύ των οποίων και διάφορες αξιολογήσεις και αναλύσεις ούτως ώστε να βελτιώσουμε την προετοιμασία των ε, προγραμμάτων και εδώ τονίζουμε για το ότι είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις αύξησης των διοικητικών ε, δυνατοτήτων για τους ε, επιλέξιμους αλλά και για τους αρχές. Πολύ σωστά είπε ο κύριος ε, Νοβακοφωτή. Είναι σημαντικό να συνεχίσει να ισχύει εγκάρσια και οριζόντια αυτό το πλαίσιο. για τη συνδιαχείριση τονίζουμε ότι χρειάζεται να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων. Αυτό βασικά είναι εθνική αρμοδιότητα με τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής και τις αξιολογήσεις. Όσον αφορά τώρα τις ε, συστάσεις όπως περιέχονται στα αποτελέσματα του ελέγχου Όλε αυτέ οι συστάσει έχουν γίνει αποδεκτέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να δούμε το πώς θα είναι βιώσιμα τα αποτελέσματα για την έγκριση των προγραμμάτων. Στην εκ των αξιολόγηση θα προσέξουμε τη βιωσιμότητα και θα εξασφαλίσουμε το ότι το νέο άρθρο 71 του CPR πρόκειται να εφαρμοστεί με ε, αυστηρότητα και πρόκειται επίσης να επιφέρουμε τις σχετικές διορθώσεις όταν δεν ε, τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Τώρα, κάτι άλλο, όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και την λογική της παρέμβασης, τονίζουμε ότι έχουμε εδώ μια σειρά στοιχείων που θα αναβαθμίσουν τον ρόλο της ε, Ελεγκτικής Επιτροπής όσον αφορά τους πόρους. Επίσης, τονίζουμε ότι οι διαχειριστικές αρχές, αλλά και οι επιλέξιμοι και οι δικαιούχοι είναι πρωταγωνιστές και σημαντικός ρόλος τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα και αλλά ο ρόλος τους θα παραμείνει ο ίδιος. Θα δούμε τι θα γίνει με τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ε, στην, στο επίπεδο του προγραμματισμού ε, περισσότερο βελληνικές για να δούμε το πώς η αξιοποίηση των ε, πόρων θα βελτιωθεί για όλους. Το σύστημα του Streamline καλύπτει τους δείκτες αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν μέσω των αξιολογήσεων με στις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτών των προγραμμάτων και της ε, πολιτικής συνοχής και της εφαρμογής της. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας παραπέμπω για άλλη μια φορά στις παραγωγές επενδύσεις που θα ε, συνεχίσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική συνοχή. θα υποστηρίζουμε τις ε, ΜΜΕ και στη συνέχεια. Για την πλευρά τη οικονομική ανάπτυξη, ο ρόλο του είναι πολύ σημαντικό και έχουν φυσικά να συμβάλλουν ε, με την οικονομική μα ευημερία. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ και για τι ε, συμπληρωματικέ πληροφορίε που δώσατε. Κύριε Μπάλκο, επιθυμείτε να λάβετε πάλι το λόγο. Μόνο για να ευχαριστήσω όλες και όλους που λάβατε το λόγο στη διάρκεια της συζητήσεως για την θετική αξιολόγηση του έργου μας. Και ευχαριστώ ιδίως τον κύριο Πυρίνσκι που έδωσε την ευκαιρία συζητήσεως τις δύο αυτές φορές που συναντηθήκαμε. Και τονίζω μόνο ότι προσωπικά εκφράζω την εικονοποίησή μου, διότι Δείξαμε σε όλους τους ενδιαφερομένους και σε εσά τους ευρωβουλευτές πως είναι σημαντικό η βιωσιμότητα να είναι σε όλη την διάρκεια του έργου. Από το σχεδιασμό μέχρι την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων κλπ. Σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου και όχι μόνο στην περιγραφή αλλά να δίνουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εσά, την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, τη δυνατότητα να διασφαλίσετε την βιωσιμότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο για την καλύτερη χρήση των ε, χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Πυρίνης και εσείς τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Η συζήτηση μόλις διεξήχθη βελτιώνει την κατανόηση του προβλήματος και δείχνει ότι έχουμε κάνει βήματα. Αφενός, η βιωσιμότητα είναι κάτι παραπάνω από την παραγωγικότητα της επένδυσης μόνο. Είναι δηλαδή μια εγκάρσια πλέον ε, ιδέα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως αποφασιστικός παράγων. Εκφράζω την εκτίμησή μου επίσης για μια δική σας παρατήρηση δηλαδή για τις πρόσθετες πληροφορίες που έδωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οφείλω ωστόσο να σημειώσω ότι δεν δείχνει πάντα την ίδια θετική στάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λάβαμε τώρα πληροφορίε και ιδίως σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό και τη λογική των παρεμβάσεων, που είναι πολύ ενδιαφέρον ως πληροφορία το streamlining, streamlining των δικτών για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι συνολικά ε, χρησιμοποίησαμε το χρόνο χρήσιμα. Ευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο βεβαίως και όλες και όλους όσοι έλαβαν τον λόγο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. ας μην κάνουμε το λάθος. Πρέπει να παραμείνουμε ιδιαίτερα απαιτητικοί απέναντι στι στις προφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι υπάρχει χώρος βελτιώσεως. Επανέρχομαι στο υπαριθμό 4, αφού τελειώσει η συζήτηση αυτού τώρα. Ο κύριος Τσέλερ είναι παρόν. Πρόκειται για την παρουσίαση του Γενικού Προϋπολογισμού της Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2019. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη μου στην Επιτροπή Αναπτύξεως όπου προβλέπονταν σημαντικές ψηφοφορίες. Εκτός τούτου και η γνωμοδότηση για το προϋπολισμό 2019. Η συζήτηση για την χορήγηση εντολής για τους τριμπηρείς διαλόγους για τον προϋπολισμό 2019 έγινε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα εκ των υστέρων συζητούμε ακόμη τις βάσεις ε, της συνολική εκθέσεως και τη γνωμοδοτήσεω. έχει καλώ. Σε λεπτομέρειε υπησέρχομαι στο σχέδιο το οποίο σας έχω υποβάλει. Για τροποποιήσει κάθετο συμπληρώσει. θα χαρώ πολύ αν μου κάνετε τέτοιες. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα γενικά είναι ότι το 2019 είναι το τελευταίο έτος Τη τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Το 2019 επίση είναι και το τελευταίο έτος της ε, Στατικής ε- Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Το 2019 είναι επίσης το τελευταίο έτος της Επιτροπής ε, της οποίας ηγείται ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Εν προκειμένου νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο της παραπέρα, της συνέχισης μάλλον των υφιστάμενων προγραμμάτων ούτως ή άλλως αυτό ε, ε, ισχύει, αλλά το έτος αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για μια γενική αναθεώρηση της στρατηγικής μας. Να μην μας συμβεί το ίδιο όπως το 2009 με τη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία απέτυχε απολύτως και δεν τη συζητεί πλέον κανείς. Να μην ξανασυμβεί το ίδιο από το 2020. Το τι θα γίνει βέβαια είναι γραμμένο στα άστρα. Έχω ρωτήσει σε διάφορες διευθύνσεις της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή, αν κάνουν σχετική δουλειά και μου είπαν όχι, τα αφήνουμε για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, χρειάζεται όμως προετοιμασία. Βλέπουμε επίσης ότι μεταξύ των ε, πιστώσεων πληρωμών που εγκρίνονται και των πιστώσεων υποχρεώσεων, η ψαλίδα ανοίγει όλο και περισσότερο. Και για τις πιστώσεις υποχρεώσεων βρισκόμαστε τώρα σε ένα ποσόν των σχεδόν 270 δισεκατομμυρίων, μιλούμε ε, για, δύο, για, για τον όγκο δύο προϋπολογισμών πιστώσεων πληρωμών. Ε, πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Έχουν γίνει οι δεσμεύσεις υποχρώσεων για διάφορα έργα που τελικώς δεν υλοποιούνται για διάφορους λόγους. Δεν μπορεί όμως αυτό να αποτελεί βάση για σωστή λειτουργία του προϋπολογισμού. Υπάρχει και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει τεθεί και στην ημερησία διάταξη λοιπόν. Διαπιστώνουμε επίσης ότι ο αριθμός των δημοσιονομικών εργαλείων αλλά και των διαφόρων καταπιστευμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά. Για τα καταπιστεύματα, trust funds δηλαδή, αναμέναμε ότι με χρήματα και του προϋπολογισμού αλλά, αλλά και με άλλα διαθέσιμα κονδύλια όπως για παράδειγμα για τη μεταναστευτική πολιτική ή για την αναπτυξιακή πολιτική, θα είχαμε δυνατότητες μόχλευσης, ώστε να συμμετάσχουν και τρίτα μέρη, και τρίτη δηλαδή, με σημαντικά ποσά. Αν δούμε τώρα όμως τα καταπιστεύματα, διαπιστώνουμε ότι οι προσδοκίες αυτές ε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν υλοποιηθεί. Η <clears throat> συμβολή από τρίτους είναι μάλλον πενιχρή και όταν καν υπάρχει ανέρχεται στο 10 15% από αυτά που διαπίστωσα. Και τότε οι χώρε μέλη που διαθέτουν τα χρήματα αυτά, γιατί συνήθως τέτοιοι είναι οι τρίτοι, πάλι μόνο υπό αιρεσιμότητα. Ο καθορισμός των στόχων που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη των οποίων διατηρείται κονδύλια του προπολογισμού και αυτά που επιτυγχάνονται ως αποτελέσματα, πάντοτε υπάρχει απόσταση. Αφενός ακούμε μηνύματα επιτυχίας σχετικά με τους ε, προκαθορισμένους στόχους, ότι δηλαδή διατίθεται κονδύλια, εκραίων κονδύλια και αυτό που γίνεται τελικά επιτόπου για τα έργα για να συμβάλλουν σε κάποια προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία τα έργα, υπάρχει, ξαναλέω, ανάμεσα στα δύο αυτά, μέγα κενό. Χρειάζεται λοιπόν ισχυρότερη συγκρισιμότητα ανάμεσα στην περιγραφή του στόχου, στη διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων και εν τέλει στην στρατηγική της εκτέλεσης επιτόπου. Κονδύλια από τα καταπιστεύματα, για παράδειγμα. Το μόνο που λειτουργεί είναι η εκροή των κονδυλίων για την εξωτερική διαχείριση των ε, trust funds και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι πάντα της τάξης του 6 με 7% και έχουν χρησιμοποιηθεί 9, 900 ε, εκατομμύρια. Κάτι όμως, αυτό όμως που συμβαίνει επί τόπου, σε ό,τι αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων, Γύρω από αυτά τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι πενιχρά. Εκεί λοιπόν πρέπει να στοχεύσουν οι προσπάθειές μας. Το άλλο μας αγαπημένο θέμα, η γεωργία δηλαδή, το έχουμε περιλάβει, 44,7% όλες οι, όλες ε, μάλλον το, ο μέσος όρος εισοδήματος ανά είναι κάτω των 4.000 ευρώ από όλες τις γεγραμμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Πρόκειται δηλαδή για πάρεργο εν τέλει. Δεν καλύπτουν με τον τρόπο αυτό οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις το κόστος επιβίωσής τους. Από την άλλη μεριά, 10% των εγγεγραμμένων δικαιούχων λαμβάνουν το 60% των κονδυλίων της κοινή αγροτικής πολιτικής που καταλήγουν σε άμεσες πληρωμές. Βλέπει κανείς και εκεί λοιπόν και αν δει κανείς και τις γέες που διαθέτουν 20% των εγγεγραμμένων αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν στην κατοχή τους το 80% των εκμεταλλευσίμων γεών. Κάτι το οποίο επιρρονεί το επιχείρημα που είπα προηγουμένω ότι δεν μπορεί παρά να απομένουν πάρα πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις οι οποίες καλύπτουν ίσα ίσα τις ανάγκες τους ή που λειτουργούν ως πάρεργο. Πρόκειται για αντίφαση που πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινιστεί και οι μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που εξαρτώνται από πληρωμές, διότι και με την αγροτική δραστηριότητα μπορεί κανείς να αποκομίσει κέρδος. Αυτό φαίνεται και από τις αυξήσεις των τιμών των γεών, όπου μια μεσαία ή μεγαλύτερη ε, αγροτική εκμετάλλευση δεν μπορεί καν να αγοράσει τα εδάφια αυτά πλέον για να επεκταθεί. Κάτι που μας ανησυχεί επίσης ακόμη είναι το ζήτημα της εφαρμογής προγραμμάτων και έργων στην πολιτική συνοχής. Επίσης τα διαθετικά ταμεία, όπου μέχρι το 2016 είχαμε, διαπιστώσαμε στην απαλλαγή του 2016 δηλαδή, ότι 7% των κονδυλίων για, είχαν απορροφηθεί για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ενώ παρέμενε ακόμα η αναγκαία επεξεργασία των υπόλοιπων δεδομένων. Για το 2017 και 2018 διαπιστώσαμε μια επιτάχυνση. Ελπίζω αυτή να συνεχιστεί το 2019. Τώρα το πώς θα επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι, αν είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανόνα νη συν 2, αυτό, και αυτό είναι γραμμένο στα άστρα. Σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές ακούω να ζητούν όλο και περισσότερα χρήματα. Από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε ότι το 2015 7 δισεκατομμύρια πληρωμών επέστρεψαν στα ταμεία των χωρών μελών. Το 2016 ήταν 10 δισεκατομμύρια πιστώσεις πληρωμών. Από τη μια μεριά λοιπόν ζητούν ενίσχυση στον, ε, στη στήλη των πληρωμών. Από την άλλη μεριά χρήματα που είχαν διατεθεί υποτίθεται για πληρωμέ, δεν απορροφήθηκαν. Και άλλη μια αντίφαση λοιπόν που θα πρέπει να συζητήσουμε. Αρκούμε σε αυτά για την ώρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, και για την επισήμανση των αντιφάσεων βεβαίως. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Εγώ μιλάω εξ ονόματος του κυρίου Μπογκάν. Έχει ζητήσει συγγνώμη γιατί έπρεπε να φύγει για να μεταβεί σε άλλη συνεδρίαση. συνάδελφος ε, ευχαριστεί τον κύριο Τσέλερ κυρίως για τις προτάσεις, ε, κάποιες προτάσεις που κάνει. Του φαίνεται θετικό το πώς ε, σκέφτεται το θέμα του να ξαναμπεί ο κανόνας νη συν και στην δυνατότητα να υπάρχει και το νη συν μας το σχολίασε και το ελεκτικό συνέδριο. Θα μπορούσαμε να γυρίσουμε σε μια μεγαλύτερη επιθαρχία... ή να πλαισιώσουμε την υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να συγχρηματοδοτήσουν. Αφού θα έχουμε περάσει το πιο κρίσιμο σημείο της κρίσης. Γιατί ξέρετε, συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα, και με προσοχή θα πρέπει να δούμε μαζί με την Κομισιόν πώς δεν θα χάσουμε την ευελιξία γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν προβλήματα Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει η ευελιξία μεν, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια πειθαρχία στον προϋπολογισμό ετησίως πρέπει να υποχρεώσουμε να εφαρμόζονται τα προγράμματα και τα κράτη-μέλη να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους έτσι όπως δεσμεύονται άπαξ 7 έτη. Ο κύριος ε, Μπογκανίλη θα ήθελε να θέσει μια ε, ερώτηση στον κύριο Τζελέρ σε σχέση με την παράγραφο 17, σε σχέση με τους δείκτες για την ε, παράτυπη μετανάστευση. Θα ήθελε να ξέρει ποιος είναι ο στόχος για τέτοιους δείκτες. Καθώς ο κύριος Τζέλερ αναφέρει την ε, αναγκαιότητα να θεσπιστούν οι δείκτες αυτοί, ποιος είναι ο στόχος λοιπόν του εισηγητή. Τι θα είναι ο στόχος των δικτών αυτών. Και για την Επιτροπή αναφέρεται ο κύριος Μπογκδάν στην παραγράφους 18 και 19 του εισηγητή. Εδώ γίνεται μια έντονη κριτική σε σχέση με τις δαπάνες ε, στο θέμα της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Και λέει ακριβώ ότι δεν ε, έχουν επισημανθεί οι δαπάνες ε, που αφορούν το μεταναστευτικό. Επομένως, αναρωτιέται ο συνάδελφος, με ποιο τρόπο μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση για τον νέο προπολογισμό. Γιατί. Εν όψη του νέου προπολογισμού θα πρέπει να πούμε με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί η ίδια κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόκειται και για ερωτήσεις προς την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών της Επιτροπής. Ορίστε, έχετε το λόγο. Η κυρία εκπρόσωπος της ε, Γενικής Διεύθυνσης. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης. Και θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια για τα κυρία σημεία. Καταρχήν, θέλω να πω ότι η Κομισιόν δεσμεύεται στο να διασφαλίσει ότι ο προπολογισμό τη Ένωση ε, θα πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα για του ε, πολίτε, διασφαλίζοντα ότι θα δίνονται οι πόροι για τι προτεραιότητε ε, και ότι κάθε δράση θα έχει προσθέμενη αξία και ψηλέ επιδόσει. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια για τους στόχους και το πλαίσιο επιδόσεων, τις ε, αποδόσεις και τα αποτελέσματα. Θέλω να τονίσω ότι η Κομισιόν συνεχίζει να εργάζεται για να βελτιώσει το περιεχόμενο των δημοσιονομικών εγγράφων της, προκειμένου να είναι ε, πιο σύντομα και πιο διαφανή και κατάλληλα εστιασμένα αλλά και βανάγνωστα. Και ήθελα να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε της ναι, επισκόπηση για τις επιδόσεις των προγραμμάτων. Αυτό αποτελεί ένα σύντομο έγγραφο επισκόπησης για τα 16 προγράμματα δαπανών. Το έγγραφο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στην ιστοσελίδα, όμως θα το τυπώσουμε ε, και θα διαναμηθεί και σύντομα στην Επιτροπή σας. Πιστεύω ότι αυτό θα διευκολύνει και την ανάλυση του κάθε προγράμματος ως ε, προς τους ε, στόχους ε, και την εφαρμογή των δικτών. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που είχε να κάνει με τη διαφορά πιστώσεων πληρωμών και πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του πολιτικού δημοσίου είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διαφορές και μάλιστα αυξάνεται και διαφορά σε αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο γιατί υπήρχαν καθυστερήσει τα πρώτα χρόνια στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι η εφαρμογή το 2017 για την πολιτική συνοχή ήταν καλύτερη από το 2016, ακόμη και αν έχουμε μειώσει τις ε, πιστώσεις, ανάληψη υποχρεώσεων, αλλά χρησιμοποιήσαμε ένα μεγάλο ποσοστό πληρωμών που ήρθαν από διορθώσεις ε, ειδικών εσόδων, εισόδων ειδικού σκοπού. Και επίσης πιστεύουμε ότι το 2018 το επίπεδο της εφαρμογής είναι καλύτερο από το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις για τη γεωργία, ότι το 20% των εκμεταλλεύσεων ε, λαμβάνει το 80% των κονδυλίων. Αυτό ο αριθμός συνοψίζει τις διαφοροποίησεις που υπάρχουν ε, στη δομή των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων. Αφενός έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων και λίγες εκμεταλλεύσεις που είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επίσης, υπάρχει και το γεγονός ότι οι πληρωμές δίνονται δυνάμει εκταρίων. Η Κομισιόν έχει εξετάσει κάποιες προτάσεις να προσπαθήσει να υπάρξει ένα ανώτατο όριο στο ποσό που δίνεται στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και στο σημερινό παλιέτες δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε ήδη προτείνει κάποια νότατα όρια που δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν για το αν θα τα εφαρμόσουν ή όχι. Όμως για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αυτά τα ανώτατα όρια θα είναι υποχρεωτικά. Η πρότασή μας για τα ανώτατα όρια θα είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη. Σε σχέση με τον κανόνα νησιν 2, νησιν 3 για τη συνοχή. Η πρόταση για το επόμενο MFF συμπεριλαμβάνει τον κανόνα νησιν 2, τον έχει επενισαγάγει η Κομισιόν. Νομίζω ότι τα κάλυψε όλα πάνω κάτω. Έχουμε και το θέμα όμως για το μεταναστευτικό, η ερώτηση της κυρίας Αγιάλα. Εμείς θέλουμε να έχουμε μία πλήρη ε, παρουσίαση όλων των δαπανών σε μία έκθεση που θα σας την παρουσιάσουμε πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο εισηγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δήλωση και για την πρόπτικη σχετικά με τις βελτιώσεις που θα επιφέρει στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και διαφορέ απόψεων και μεταξύ των συναδέλφων, αν και ίσως εδώ όχι τόσο πολύ, στην παρουσία επιτροπή δηλαδή. Εάν για τη γνωμοδότηση του 2019 έχουν οι συνάδελφοι μου ακόμα τροπολογίε ή συμπληρώσει. ευχαρίστω. Κάτι το οποίο περιέλαβα και το δηλώνω ρητά είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου στην έκθεση λέμε ότι πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς και σε ό,τι αφορά το προσωπικό, αλλά βεβαίως και να εξοπλιστεί επαρκώς, με επαρκή εξοπλισμό. Διότι τα όσα έχουν προταθεί ως τώρα μας φαίνονται υπερβολικά περιορισμένα. Το τονίζω αυτό, λέει η Πρόεδρος, όπως φαίνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την προκοδότηση που της έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τώρα, μάλλον θα είναι θνησιγενής. Θα καταλήξουμε σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας. Και οφείλω και εγώ λοιπόν να προειδοποιήσω. Αναμένουμε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Επιτροπής για τα πολιετή προγράμματα, την ανάλυση, το οποίο θα συζητήσουμε. Μάλλον εγώ το έχω διαβάσει ήδη. Έχω και κάποιες αμφιβολίες για το αν είναι το σωστό, διότι σε ορισμένα πράγματα καταλήγεται σε θεμελιωδώς διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που έχουμε από το ελεγκτικό συνέδριο. Θα αναλύσουμε ωστόσο την αξιολόγηση αυτή πάρα πολύ προσεκτικά. Η κυρία Σέντερ πάλι. Για τον κύριο Μπόκαν θέλω να πάνω μπορεί να πει κάτι την παράγραφο 17 εκεί που λέει ότι θα πρέπει να έχουμε θέσπιση κάποιων ε, δικτών και να απαλληφθούν αυτές οι αιτίε που αφορούν την παράνομη μετανάστευση. Και θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο έχουμε εδώ αυτούς τους δείκτες. Γιατί είναι κάτι ευρύτερο αυτές οι αιτίε που λέμε να απαλληφθούν. Αν μπορείτε να μας τα πείτε. Η κυρία Μπουσκές. Uh, Αυτοί οι δείκτες που αφορούν την μετανάστευση θα το δούμε σχετικά με αυτούς με την DG Home. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω τώρα περισσότερο. Το μόνο που μπορώ να σας πω από τώρα ότι αυτά αφορούν την ε, ευρύτερη έκθεση για την μετανάστευση. Ο κύριος Τσέλερ, ε, ας κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην καταπολέμηση των αιτίων της μετανάστευσης, εκεί πιο πολύ είναι ζήτημα πολιτικής της ανάπτυξης, γειτονίας. Αυτό που τίθεται στο προσκήνιο εδώ, εν προκειμένου στη γνωμοδότηση, είναι η πολιτική ενσωμάτωσης ή ένταξης. Η υποστήριξη της πολιτικής ενσωμάτωσης των χωρών μελών, όπου πρόσφυγες ή και μετανάστες έχουν καταλήξει, έχουν φτάσει δηλαδή. Εδώ είναι προκειμένο... σε ό,τι αφορά τάξη μεγέθους των ανθρώπων που έρχουν, έρχονται στην Ευρώπη, δεν είχε προβληθεί τίποτα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά και στου εθνικούς προπολογισμού εξ όσων γνωρίζω, αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι και στα τελευταία δημοσιονομικά έτη είχαν πάρει χρήματα από διάφορα κονδύλια των προπολογισμών για να προσφέρουν στήριξη στις χώρε μέλη από το ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποδοχή μεταναστών ή για προγράμματα ενταξή τους. Τώρα πάμε να φτιάξουμε ειδική προσέγγιση και θα ήθελα να γνωρίζω, εάν υπάρξει, αν διατυπωθεί δηλαδή ειδική προσέγγιση του προπολισμού, ποια πράγματα θα χρηματοδοτούνται, με ποιου στόχου και αν υπάρχουν μετρήσιμοι και συγκρίσιμοι δείκτες σύμφωνα με τους οποίους κατανέμονται τα κονδύλια αυτά. Ή γίνεται στη βάση της αρχής όποιος φωνάζει περισσότερο παίρνει περισσότερα μιλώ για δαπάνες καταλήμματων, ε, ε, καταλήματον ε, εκπαίδευσης, υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Άλλωστε, στην κοινωνική πολιτική έχουμε αρχίσει και υιοθετούμε δείκτες για τη μέτρηση της απόδοσης της κοινωνικής πολιτικής, τουλάχιστον από τη Γερμανία αυτό γνωρίζω, ώστε στην απόδοση λογαριασμών να είναι σαφές περί τίνος πρόκειται. Έτσι το σκέφτομαι αυτό τώρα. Εάν δηλαδή υπάρξει μακροπρόθεσμη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών η Σας ευχαριστώ. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 6 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, 14 μάλλον. Συνεχίζουμε τώρα με σύντομες παρουσιάσεις ειδικών εκθέσεων για βελτίωση της νομοθεσίας η 16-2018 επειδή ο κύριος Γκρέτεν κολλείεται σήμερα θα αναλάβει την παρουσίαση της εκθέσεως ο επικεφαλής του ιδιωτέρου γραφείου του, κ. Όστερτ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρώτα-πρώτα παρακαλώ συγχωρήστε τον κύριο Άρη Κρέτεν που είναι ο εισηγητής για αυτή την δική έκθεση. Δεν μπόρεσε να έρθει εδώ ο ίδιος, έπρεπε να μείνει στο Λουξεμβούργο για να συμμετάσχει σε σημαντική συνάντηση του Ελληνικού Συνεδρίου για να υπάρξει η απαρτία. Οπότε μου έκανε την τιμή να μου αναθέσω να τον εκπροσωπήσω κύριε και κύριοι. Αυτή η ειδική έκθεση που σήμερα σας παρουσιάζουμε αφορά το, την εκ των υστέρων αξιολόγηση αυτής της υπόθεση τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωσης που ονομάζεται για μια καλύτερη νομοθεσία Ούτω ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους ε, διάφορους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κατά αυτό το έργο μας εξετάσαμε εάν αυτές οι διαδικασίες που προβλέπονται έχουν προγραμματιστεί σωστά, εάν έχουν εκτελεστεί σωστά, εάν έχουν ε, περάσει από την σωστή διαχείριση και έλεγχο ποιοτικό, ε, ώστε να βελτιωθεί η νομοθεσία. Θα πρέπει να δούμε ακριβώ ποιο είναι το βελενικέ αυτού του ελέγχου που αφορά δύο διαφορετικά σημεία. Πρώτα-πρώτα ε, την επαναξιολόγηση εκ των υστέρων τη ε, νομοθεσία, τη περίοδου 2013 μέχρι το 2016 και για τέσσερις γενικές διευθύνσει τη επιτροπή DG Home, Santé, Grow και Env, περιβάλλον δηλαδή. Και επίσης ε, αυτό αφορά το σύνολο των νομοθετικών πράξεων και επίσης των αναλύσεων, επιπτώσεων εκ των προτέρων όπως ε, εγκρίθηκαν μεταξύ του 2014 και 2016. Πρώτα-πρώτα είπαμε να δούμε σε ποιο βαθμό η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έλαβαν υπόψη αυτές τις σχετικές ρήτρε για επανεξέταση και παρακολούθηση οι οποίες προβλεπόντουσαν δεύτερο να δούμε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήρησε όλες τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την εκ των υστέρων επανεξέτηση και επίσης όσον αφορά τις κανθυντήριες γραμμές, τα πρότυπα και τους μηχανισμούς ελέγχου ποιότητος τρίτων, να δούμε αν η Επιτροπή και οι συνομοθέτες ε, εξασφάλισαν ότι υπήρξε δημοσιοποίηση αυτών των ε, αξιολογήσεων και κατά πόσον υπήρξε παρακολούθηση ε, της ε, εξέλιξης όσον αφορά τον ε, νομοθετικό κύκλο. Τέταρτον, να δούμε το κατά πόσον είχε σωστά περιχαρακωθεί το πρόγραμμα REFIT, για να δούμε τώρα κατά πόσον υπήρξε συμβολή από όλη αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη νομοθεσία. Πριν απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, πρέπει να σταθούμε στο ότι το Ελληνικό Συνέδριο θεωρεί ότι αυτό το σύστημα της επαναξιολόγησης ε, ε, την χάνει αποδοχής από τα κράτη-μέλη. Για να δούμε τώρα. Έχει ένα σύστημα καλής διαχείρισης και έλεγχο ποιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βοηθά αυτό στην ε, βελτίωση της νομοθεσίας. Όμως, επίσης, έχουμε επισημάνει κάποια αδύνατα σημεία. Δηλαδή, συγκεκριμένα, πρώτα-πρώτα, ε, διαπίστωσαν οι ε, πάρεδροι του συνεδρίου το ότι υπήρξαν αυτές οι ρήτρες οι οποίες ε, υπήρχαν στην νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε ότι δεν υπήρξαν διοργανικές κατευθυντήριες γραμμές. Οπότε το περιεχόμενο αυτών των ρητρών επαναξιολόγησης και τα αποτελέσματα ε, δεν ήταν πάντοτε ξεκάθαρα δεύτερον. Είπαμε ότι αυτή η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τις προκθέσεις που τάσσει ο νόμος, η καλή πρακτική, οπότε είπαμε ότι δεν έχουμε ε, άρα τελικά μια αξιολόγηση ε, με τη στενή της έννοια. Οπότε οι καθημερινές γραμμές δεν εφαρμόστηκαν παρά μόνο από το 2017. Τρίτη παρατήρηση ε, διαπίστωσε το συνέδριο ότι όλα αυτά τα σχετικά έγγραφα υπήρχαν προσβάσιμα στο κοινό. Τα περισσότερα από αυτά ε, ήταν ε, ξεκάθαρο το τι μέτρα αφορούσαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά διεβίβαζε εκ των υστέρων στους συνομοθέτες όλα αυτά τα έγγραφα σε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Ε, όμως, τελικά το Συμβούλιο δεν είχε αντιδράσει σε αυτήν ε, την επικοινωνία. Το Refit επίση είπαμε ότι δεν ήταν σαφές ποια ήταν τα κριτήρια ούτω ώστε κάποιες πρωτοβουλίες να καλυφθούν από το Refit. Κυρίες και κύριοι, επί τη βάση όλων αυτών των διαπιστώσεων έχουμε ε, να προτείνουμε τα εξής. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον και πιο σημαντικό, θα πρέπει να θωρακίσει τη διοργανική συμφωνία που ονομάζεται καλύτερη νομοθεσία σε συνεργασία με Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και στα πλαίσια της ισχύου της διοργανικής θα πρέπει να επεξεργαστεί ένα εγκόλπιο διοργανικό όσον αφορά τις ρήτρες επαναξιολόγηση. Χρειάζεται επίση κάποιο κατάταξη των διαφορετικών ειδών ε, αποτελεσμάτων επαναξιολογήσεων ex post. Ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν κάποιοι προσανατολισμοί και ένα ενδεικτικό καλαντάρι για κάθε είδους τέτοια επαναξιολόγηση. Ε, ε, το ίδιο αφορά και κάποιες άλλες ε, ρήτρε της ελέγχου παρακολούθησης και θα πρέπει σύμφωνα με το 295 της συνθήκης να αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά πώς είναι δυνατόν να υπάρξει μια καλύτερη διοργανική συμφωνία για αυτή την νομοθεσία. Δεύτερη ε, σύσταση. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η καλύτερη ε, ποιότητα των επαναξιολογήσεων εξ post και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει κάποιους ελάχιστους κανόνες για την επαναξιολόγηση ε, πέραν των αξιολογήσεων και έτσι να υπάρχει εγγύηση ποιότητα σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία να διευρύνει το δικαίωμα ελέγχου της Επιτροπής Ελέγχου πέραν των αξιολογήσεων και θα πρέπει με τέτοιου είδους ελάχιστους κανόνες για την ποιότητα ε, μέσω των επαναξιολογήσεων να προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής ε, κατά λεπτός ποια της, της, της μεθοδολογίας της χρησιμοποιουμένης και ε, θα πρέπει να καθορίζονται τα όρια αυτών των ενεργειών κατά λεπτός, να αναλυθούν τα παραθυράκια και επίσης οι δυνατότητες διαχείρισης και θα πρέπει στο καταλληλό επίπεδο να αναλύει ποια είναι τα, τα παράθυρα, τα κενά, να υπάρχουν τα δεδομένα που χρειάζονται για τις επαναξιολογήσεις ex post και ε, κατόπιν να λαμβάνονται τα απαραίτητα δέοντα μέτρα θα πρέπει να ισχύει η αρχή ε, αξιολόγηση πριν ανάληψη ενεργειών, ούτω ώστε θα ε, συστηματικά να ισχύει αυτή η αρχή στα πλαίσια ε, κάποιου νομοθετήματος να αξιολογήσει τις επιπτώσεις κάποιας προτάσεως επί τη βάση των προηγουμένων αξιολογήσεων θα πρέπει κάθε χρόνο να, ε, αναφέρει ποιες είναι οι αναλύσεις επιπτώσεων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Το REFIT να ληφθεί υπόψη σε αυτή την προσπάθεια βελτίωσης της νομοθεσίας και θα πρέπει το REFIT να έχει πρωταγωνιστικό ε, ρόλο και να μην δίνει την εντύπωση ότι είναι κάτι το διαφορετικό από τη συνήθεια διαδικασία βουλτής νομοθεσίας. Και σας ευχαριστούμε κύριε και κύριοι, όσον και σας προτείνουμε να υλοποιήσετε αυτές τις συστάσεις. Ευχαριστώ. Το λόγο δίνω στον κύριο Χέις που είναι ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ούτε με Ως ε, εισηγητής για την γνωμοδότηση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του σε σχέση με την εξωτερική θεώρηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη η έκθεση και αν ε, δούμε την ιεράρχηση προτεραιοτήτων αυτή της Κομισιόν ε, όλου του θεματολογίου για την καλύτερη νομοθεσία, αυτό ήταν ένα κύριο θέμα της Κομισιόν να προσπαθήσει να πετύχει αποτελέσματα στον τομέα. Γιατί για τον καθημερινό πολίτη ε, πρόκειται για μείωση του κόστους ε, της νομοθεσίας ε, και για διασφάλιση ότι υπάρχουν πραγματικά ωφέλη στην προσέγγιση που θετούμε σε αυτό το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτες με το Συμβούλιο. Επομένως, ε, πάντοτε πρέπει να ρωτάμε γιατί έχουμε αυτή την νομοθεσία, μας ωφελεί και θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε στους πολίτες ε, ξεκάθαρα σε σχέση με τα ωφέλη της νομοθεσίας και από τις αναθεωρήσεις ε, που ακολουθούν ε, γιατί εμείς ε, εδώ έχουμε εγκρίνει κάποιες αναθεωρήσεις όμως νομίζω ότι η διαδικασία της ε, επισκόπησης είναι πάρα πολύ σημαντική. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έκθεση του λεκτικού Συνεδρίου και το συγχαίρουμε για το έργο του. Το γεγονός ότι είναι ένας ευρύς έλεγχος σε μία τριετή περίοδο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπως ήδη υπόθηκε, συμμετείχαν τέσσερις γενικές διευθύνσεις, Grow, Homes and Envy. Και η έκθεση περιγράφει το σύστημα σε σχέση με τις αξιολογήσεις και ποια ήταν η διαχείριση. Όμως, σε ό,τι αφορά τις ε, επισκοπήσεις, ε, υπάρχουν κάποιες αδυναμίες ε, στο σύστημα η έλλειψη κοινών κατευθυντηρίων γραμμών ε, για τις ε, αναθεωρήσεις και παρακολούθηση είναι ένα ξεκάθαρο ζήτημα. Είχαμε και την περίπτωση ότι το 2017 ε, μόλις μπορέσαμε να θεσπίσουμε μια εργαλειοθήκη για την καλύτερη νομοθεσία, όμως χρειάστηκε χρόνος και φυσικά υπήρχε πρόβλημα στο παρελθόν που δεν υπήρχε και υπάρχουν και κάποια ζητήματα σε σχέση με τα επαρκή, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα που φυσικά αφορούν οποιοδήποτε εκ των υστέρων αναθεώρηση. Επίση, και το θέμα τη βελτίωση τη συλλογή των δεδομένων και το ότι ε, πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσει γιατί καθυστέρησαν οι εξ των υστέρων αναθεωρήσεις. Αν βάλουμε κάτι στην πρωτογενή νομοθεσία και περιμένουμε να συμβεί και δεν συμβαίνει, γιατί το κοινοβούλιο δεν, στο κοινοβούλιο δεν έχει εξηγηθεί γιατί ε, δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό που κάναμε στην έκθεση είναι ότι δίνουμε κάποιες συστάσεις. Καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Ελεκτικό Συνέδριο για τις συστάσεις και τις ε, υιοθετώ. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι η Διοργανική Συμφωνία για την Καλύτερη Νομοθεσία το 2018 θα έχουμε ένα πλαίσιο και κυρίως ε, για το εγχείρημα τη παρακολούθηση και ξέρω ότι αργότερα φέτο ε, θα έχουμε και μία διοργανική συνάντηση υψηλού επίπεδου που θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Αυτό το καλωσορίζω και θέλουμε να το κάνουμε αυτό σε πιο τακτική βάση. Τρίτον, Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι καλό το μέγεθο του ελέγκτου και η ανάπτυξη περαιτέρω δικτών για να παρακολουθηθεί η εφαρμογή τη συμφωνία. Αυτό θα είναι κάτι ζωτικό καθώς το προχωρούμε για να διασφαλίσουμε ότι ισχύει η συμφωνία και λειτουργεί για όλε τι πλευρέ. Τέταρτον, πιστεύω ότι η ενεργή συμμετοχή του ελεκτικού συνεδρίου πρέπει να συνεχιστεί στον τομέα αυτό. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη όπως αναφέρω και στην νομοδοτησή μου, αλλά και το γεγονός ότι μπορούν ε, να παρακολουθούν αυτό το τομέα θα προσφέρει μεγαλύτερα ωφέλη ε, σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Έτσι λοιπόν από τη σκοπιά της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε την συνεχιζόμενη συμμετοχή του, του ελεγκτικού συνεδρίου στον τομέα. Επίσης, οι κοινέ κατευθυντήριες γραμμές για τις αναθρήσεις ε, ex post θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι διάφορε προσεγγίσει και για το λειτουργούν αυτέ οι κατευθυντήριε γραμμέ. Και τέλο, ένα πολύ σημαντικό τομέα είναι το θέμα του ενιαίου πλαισίου για τη μεταφορά στο δίκαιο των κρατών μελών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν υπάρχει μία και μόνη προσέγγιση σε σχέση με το πώ μεταφέρουν στο ιστορικό του δίκαιο τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με έναν αποτελεσματικό ω προ το χρόνο τρόπο. Και νομίζω ότι ένα ενίο πλαίσιο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ζητάμε ε, χωρίς ενοχές. Αν ε, ε, θέλουμε να έχουμε ικανή ευρωπαϊκή νομοθεσία και υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να υπάρχει και μια λογική μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο με αποτελεσματικό τρόπο, αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εργαστούμε στο μέλλον. Και η έκθεση αυτή είναι μια ευκαιρία να το τονίσουμε. Και αυτό το έχω πει και εγώ και στις δικές μου συστάσεις. Θα ήθελα να ακούσω και τις απόψει των άλλων συναδέλφων. Συγχαρητήρια και στο λεκτικό συνέδριο για την πολύ καλή δουλειά. Κυρία Γιάλα, ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, λυπάμαι που δεν είναι εδώ αρμόδιος συνάδελφος ε, από το ελεκτικό συνέδριο. Πάντως πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι θα πρέπει να είναι εδώ αρμόδιος. Τώρα υποστηρίζω πλήρω όσα έκανε ο κ. Χέης προς την ποιότητα της έκθεσης. Μας δίνει ένα δυναμικό όραμα για κάτι που για μας ήταν θεμελιώδη και πρόκειτο και για μία από τις μάχες που δώσαμε απέναντι στο Συμβούλιο. Αν και συμφωνούσαμε και πάντοτε υποστηρίζαμε την στρατηγική της καλύτερης νομοθεσίας, ακριβώς για να έχουμε μια ταχύτερη και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων που υιοθετούμε, συζητούμε και τροποποιούμε σε αυτό τον οίκο. Μου φαίνεται παρόλα αυτά ότι στο Refit κάποια στιγμή δεν εισακούστηκε υπαρκώς στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή ότι πρέπει να ενισχυθεί η εκ των υστέρων αναθεώρηση και ότι αυτό πρέπει να είναι δεσμευτικό τμήμα μιας διοργανικής συμφωνίας. Επίσης μου φαίνεται πολύ σημαντική η πρόταση για το ενίο πλαίσιο για τη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο της νομοθεσία. Γιατί δημιουργούμε μεγαλύτερα προβλήματα και στη χώρα μου υπάρχει τεράστια καθυστέρηση της ε, μεταφοράς στο ιστορικό δίκαιο ορισμένων οδηγιών. Συσσωρεύονται δηλαδή διάφορες ε, απογοητεύσεις ε, <laughs> και σε επίπεδο κυβέρνηση αλλά και σε επίπεδο πολιτών. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου αν στη μελέτη αυτή μπορέσατε να προσδιορίσετε σε ποιο βαθμό Ουσιαστικά το Συμβούλιο διευκολύνθηκε για να αποσύρει κάποιους φακέλους που ενδιέφεραν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς είχαμε εργαστεί επί αυτών ε, των φακέλων και είχαν μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο και με όλη αυτή τη διαδικασία του Refit ε, δεν χρειάστηκε να αναλάβει καμία δέσμευση το Συμβούλιο. θέλαμε να μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοια προβλήματα γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε και αυτή την εικόνα. Δηλαδή για το θέμα της διοργανικής ισορροπίας, σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχουμε επαρκή ε, ε, αρμοδιότητα ανάληψης πρωτοβουλίας εδώ στο Κοινοβούλιο. Και επομένως αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε και ένα είδος περιορισμού της εντολής μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάτσον από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορίστε. this one working? Yes. Φαίνεται πως αυτό το μικρόφωνο λειτουργεί καλά. Με συγχωρείτε, λέει ο κ. Σουάτσον. Όπως έλεγα, λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Χώστερτ για την παρουσίαση, καθώς και τον κύριο Χέις για την ε, παρέμβασή του και τους άλλους συναδέλφους σας για τις απόψεις που εξέφρασαν. Πρόκειται για έκθεση που εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουμε με πολύ ευνοϊκό ε, πνεύμα και γενικά θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε καλύτερα τον τρόπο, τρόπο σκέψεώς μας και βελτιώσεως των αξιολογήσεων. Και ένα βασικό μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι η βελτίωση της νομοθεσίας είναι και μια διαδικασία μάθησης για μας. Αναζητούμε διαρκώς βελτιώσεις για το πώς θα τα καταφέρουμε καλύτερα και η έκθεση που παρουσίασε ο κ. Χώστερτ είναι σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι πέραν αυτού της, της γενικής τοποθετήσεως υπάρχουν δύο πτυχές της εκθέσεως που μας ικανοποιούν πολύ. Αφενός, ότι δείχνει καθαρά ότι είναι ε, βασική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογεί την νομοθεσία της και τα προγράμματά της. Υπάρχει όμως και ε, ισχυρό διαθεσμικό ε, στοιχείο. Μπορεί να επιτύχει η βελτίωση νομοθεσίας μόνο εάν συνεργαστούν στενά τα τρία θεσμικά όργανα ώστε η νομοθεσία που στείλουμε στα πόδια της πραγματικά να εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα το οποίο ε, βγαίνει από την έκθεση αυτή. Το δεύτερο που ε, βρίσκομαι ε, σωστό είναι η αναγνώριση ότι σε σύγκριση με τις χώρες μέλη και στην βάση διεθνών συγκρίσεων τα καταφέρνουμε αρκετά καλά. Αυτό μάλιστα στην βάση εργασιών του ΟΟΣΑ ε, για το ρυθμιστικό πλαίσιο ε, του 2015. Ο ΣΑ συντάσσει ε, νέα νομοθετική προοπτική για τα τέλη του τρέχοντος έτους και νομίζω ότι θα τα πάμε καλύτερα εκεί, στις κρίσεις δηλαδή του ΩΣΑ, από ό,τι το 2015. Αντιλαμβανόμαστε ότι για όλες τις πτυχές βελτίωσης της νομοθεσίας όπως είπα, είναι μια διαδικασία μάθησης και παρόλο που τα πάμε καλά σε σύγκριση με τις χώρες μέλη αλλά και διεθνώς, παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα πολύ περιθώριο βελτιώσεως. Θα δώσουμε συνέχεια σε όλες τις συστάσεις που έχει θέσει υπόψη μας το ελεγκτικό συνέδριο, είτε πλήρως είτε εν μέρη, αυτό εξαρτάται από την επιμέρους σύσταση. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ σε μια ή δυο από τις συστάσεις αυτές. Η πρώτη σύσταση που σωστά υπογραμμίζει ο κύριος Χώστερ το ότι έχει κέρια σημασία είναι αυτή που αναφέρεται στην διαθεσμική πτυχή του θέματος. Και σε ό,τι αφορά τις ε, κοινέ κατευθυντήριες γραμμές για την εκ των υστέρων επανεξέταση. Εμεί, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστώ, θα συνεργαστούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα, με τα δύο άλλα θεσμικά όργανα, για την σύνταξη αυτών των κατευθυντήριων γραμμών στη βάση των όσων έχουμε ήδη επιτάπητος, χωρίς βεβαίω να λέμε ότι είναι και το τελικό προϊόν, διότι θα πρέπει να εγκριθεί και από τα τρία θεσμικά όργανα. Αντιλαμβανόμαστε ότι εξαρτώμεθα από τα δύο άλλα θεσμικά όργανα και θεωρούμε ότι και το Συμβούλιο στην απάντησή του στον έλεγχο ίσω να μην φανεί τόσο ενθουσιώδε όσο εμείς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η αντίδραση του Συμβουλίου και θα πρέπει να την εντάξουμε και αυτήν στο διαθεσμικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την συλλογή των δεδομένων που αναφέρει ο εισηγητής, και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι έχει κρίσιμη σημασία ότι η διαθεσιμότητα σωστών δεδομένων, επίκαιρων δεδομένων είναι απολύτω αναγκαία για την βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεών μας. Και αυτό απηχείται άλλωστε και στη Διαθεσμική Συμφωνία για Βελτίωση της Νομοθεσίας. Πάλι λέγω ότι αποτελεί βασική ευθύνη των χωρών μελών όταν συνεργάζονται μαζί μας να φροντίζουν να διαθέτουν τα σχετικά δεδομένα. Εμείς πάντως εργαζόμαστε και εσωτερικά και νομίζω η εσωτερική αυτή εργασία έχει λάβει σημαντική όθηση με τις πρόσφατες ε, ρυθμίσεις για το, για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα δεδομένα αυτά όταν δεν είναι διαθέσιμα θα πρέπει να ε, δούμε πώς θα μπορούμε να τα συλλέγουμε. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά για μας. Εν τέλει και σε ό,τι αφορά το REFIT, εδώ έχουμε μια σχετική διαφορά απόψεων με το ελεγκτικό συνέδριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια έννοια η οποία έχει εξελιχθεί μέσα στον χρόνο και ότι στις αρχικές τη φάσεις ίσω να μην ήταν τόσο σαφή, ή τόσο στοχευμένη όσο θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι σύν τον χρόνο έχουμε κατορθώσει να τα διευκρινίσουμε τα πράγματα αυτά και να δημιουργήσουμε με το πρόγραμμα Refit και με την πλατφόρμα Refit ένα ας πούμε σήμα κατατεθέν το οποίο είναι γνωστό, έχει γίνει αντιληπτό και ε, στα πλαίσια όχι μόνο πλέον των επιχειρήσεων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη μείωση των επιβαρύνσεων και για τις άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές που πάντοτε εκφράζουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ανησυχία, αντιλαμβάνονται ότι κάνουμε την προσπάθεια να μειώσουμε την επιβάρυνση, χωρίς όμως να θίγουμε τους βασικούς στόχους της πολιτικής μας. Το REFIT λοιπόν ως σήμα έχει γίνει ε, καλά αποδεκτό και κατανοητό από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βεβαίω, σύμφωνα με τι συστάσει του Ελεκτικού Συνεδρίου, θα βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω την προσέγγιση αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν θα δώσω σε κανέναν άλλο το λόγο, διότι πρόκειται για σύντομη παρουσίαση. Εδώ λίγη λοιπόν η συζήτηση του θέματο αυτού. Συνεχίζουμε με σύντομη παρουσίαση του ενημερωτικού εγγράφου του Ελεκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απλούστευση τη άσκηση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Ε, δίνω 15 λεπτά για όλο το εγχείρημα αυτό, οπότε δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Μπάλκο. Θα ξεκινήσω. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, κυρίε κυρίε και κύριοι, ο στόχο αυτού του εγγράφου είναι να συνεισφέρει στην προετοιμασία του νομοθετικού πακέτου και στη συζήτηση τη της ε, τη ε, πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Παρουσιάζουμε τέσσερις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που θεωρούμε σημαντικές για τη διαδικασία της απλούστευσης και πέντε κύριους τομείς για αποτελεσματική απλούστευση. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η παράδοση της παραδοσιακής πολιτικής έχει γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη. Παρ' όλα αυτά η πρώτη αρχή που έχουμε εντοπίσει είναι η ανάγκη για μια καλά προσδιορισμένη στρατηγική. ανάλυση μας ε, των απόψεων των ε, διάφορων πρωταγωνιστών, όπως βλέπετε στο κεκτημένα του εγγράφου μας δείχνει ότι δεν υπάρχει γενική συμφωνία για τους στόχους της απλούστευσης και γι' αυτό ε, δηλαδή για ποιον και πώς απλοποιούμε. Ένας από τους κύριους στόχους της διοικητικής απλούστευσης είναι να αφαιρεθεί το ε, μη απαραίτητο κόστος, μειώνοντας το διοικητικό άχθος για τους δικαιούχους και τις ε, αρχές των κρατών μελών. Η απλούστευση θα πρέπει να συνάδει με αυξημένη αστεία στις επιδόσεις, την αποτελεσματικότητα του κόστους και ποιοτική ρύθμιση. δεύτερη αρχή καλή για μια διορθωμένη προσέγγιση βάση αποδείξεων για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα και να προτείνουμε την απλούστευση. Οποιαδήποτε πρόταση απλούστευση θα πρέπει να βασίζεται σε εύρωστε αποδείξει για να μεστρεθεί ο κινδύνο ότι η απλούστευση μπορεί να επικεντρωθεί σε δραστηριότητε ε, που ε, ουσιαστικά μπορεί να ενοχλούν ε, τα υποκείμενα, αλλά ίσως να μην είναι πιο επαχθή. Στο ε, σημείο θα πρέπει να είναι μία πλήρης επισκόπηση της προέλευσης του βάρους στα επιχειρησιακά προγράμματα και ο εντοπισμό των μη απαραίτητων κόστος και της μη απαραίτητης πολυπλοκότητας. Μία σημαντική πολύ πολυπλοκότητα για τους δικαιούχους είναι ο κανονιστικός υπερθεματισμός, δηλαδή απαιτήσει ε, που έχουμε σε εθνικό επίπεδο πέρα από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προκύπτουν από έλλειψη ασφαλείας δικαίου και τι ανησυχία ότι μία λιγότερη αυστηρή ερμηνεία των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχουν αποτέλεσμα να επιβάλλει η Κομισιόν δημοσιονομικέ διορθώσει. Η απλούστευση δεν θα πλέπει μόνο να βασίσει στι αποδείξει, αλλά να είναι και διαρθρωμένη, δηλαδή εντοπισμό και ποσοτικοποίηση του άχθου, ε, εξάντε μελέτη αντικτύπου και εξάρτητο έλεγχο και θέσπιση στόχων για τη μείωση του άχθου και ε, παρακολούθηση τη διαδικασία. Η πραγματική απλούστευση χρήζει δέσμευση από όλου του παίκτε, την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην πρόταση, διαπραγμάτευση και υιοθέτηση του νομικού πλαισίου, αλλά και των κρατών μελών, καθώ θέτουν του κανόνε για του δικαιούχου, ε, για την επιλογή των ε, επιχειρήσεων, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτούς και συνεισφέρουν ε, στο διοικητικό άχθος. Το τέταρτο αφορά τη λογοδοσία και τις επιδόσεις. Η απλούστευση δεν είναι αυτός ο σκοπός και δεν θα πρέπει να διακυβεύει τα επιτεύγματα ε, στους ενισχυμένους εσωτερικούς ελέγχους. Ε, η δουλειά μας μας δείχνει ότι κάποιες ισχυρές διευθετήσεις λογοδοσίας συνεισέσφεραν σε σημαντική μείωση στο επίπεδο των παρατηρήσεων τα επιτεύγματα αυτά δεν θα μπορούσαν να είναι δυνατά χωρίς ενισχυμένους ελέγχους και δεν θα πρέπει να δικηδευτούν από την απλούστευση εις βάρος της λογοδοσίας για τη χρήση δημοσίων κονδυλίων. Επίσης, η απλούστευση θα πρέπει να συνάδει με αυξημένη εστίαση στις επιδόσεις, γιατί είδαμε ότι η έλλειψη εστίαση στις επιδόσεις είναι ένα κύριο πρόβλημα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τώρα, θέλω να αναφερθώ στους πέντε τομείς κλειδιά για την απλούστευση της πολιτικής ο πρώτο τομέα είναι η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η καθοδήγηση. Η απλούστευση ξεκινά με απλού, ε, σαφεί και σταθερού κανόνε και με μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων που σχετίζονται με τα διάφορα κονδύλια και προγράμματα. Μεταξύ των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων ο αριθμός ε, των σελίδων των κανονισμών ε, διπλασιάστηκε από 1732 σε 3889. Και λόγω των ε, καθυστερήσεων της υιοθέτησης του νομοθετικού παχέτου για τη συνεχή για τη σημερινή προγραμματική περίοδο, τονίζουμε τη σημασία ε, του να έχουμε τους κανόνες εγκαίρως ε, καθώς και τη σταθερότητα των κανόνων κατά τη διάρκεια και μεταξύ των προγραμματικών ε, περιόδων. Επίσης, οι σταθεροί κανόνες σημαίνουν αποτελεσματική απλούστευση και κάποιες αλλαγές στο σημερινό σύστημα θα μπορούσαν να καταφερθούν κατά των πρόσφατων επιτευγμάτων στη βελτίωση της νομιμότητας και της κανονικότητας της πολιτικής συνοχής. Η απλούστευση δεν αφορά μόνο τη σύντμηση των κανόνων και τη ε, μείωση ε, του συνολικού αριθμού του. Αυτή είναι ποσοτική απλούστευση, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ποιοτική απλούστευση. Δηλαδή, οι κανόνες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό. Ο δεύτερος τομέας κλειδί είναι η ε, διαχείριση η δομή διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Έχουμε περίπου 1.400 αρχές ε, διαχειριστικές ε, ε, για πάνω από 390 επιχειρησιακά προγράμματα στα κράτη-μέλη, καθώς υπάρχει μεγάλη αυτονομία. Αυτό αποτελεί πρόκληση για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ο των προγραμμάτων, των αρμόδιων αρχών, αλλά και των εξάντε όρων τις εξάντερες και του πολύ μεγάλου αριθμού των ε, δικτών επιδόσεων ε, είναι κάτι σημαντικό. Τρίτος ε, στόχος έχει να κάνει με την απλούστευση της επιλογής των σχεδίων και της εφαρμογής και αντιμετωπίζοντας και την κανονιστική υπαρθεματικότητα. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός σχεδίων που θα μπορούσαν να εποφεληθούν από τη χρήση των καλύτερων τεχνολογιών. Αναφέρομαι στο παράδειγμα 3 του εγγράφου ε, που μας δείχνει ότι πολλές διαφορές υπάρχουν σε σχέση με το πώς κατατίθενται οι αιτήσει και το μεγεθός τους. Ο τέταρτος τομέας για την απλούστευση είναι η χρήση ε, των ε, επιλογών απλουστευμένων κόστος. Αυτό μπορεί να μειώσει το διοικητικό άχθος για τους δικαιούχους και να βοηθήσει να μειώσει το κόστος της εφαρμογή. και στην ε, σημερινή περίοδο ήταν το μέτρο που χρησιμοποιήθηκε περισσότερα. Ο κανονισμός Omnibus, ε, το σχέδιο του κανονισμού διευρύνει το πεδίο εφαρμογή ε, και την εφαρμοσικομότητα αυτών των επιλογών απλουστευμένου κόστος. Οι αναθεωρήσεις του Omnibus αν υιοθετηθούν θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του διοικητικού άχθους. Ο πέμπτος τομέας για την απλούστευση σχετίζεται σε πιο αποτελεσματικούς ελέγχους όπου οι επαληθεύσεις της διαχείρισης από τις διαχειριστικές αρχές και τους φορείς ε, καλύπτουν την πλειοψηφία. Η εμπειρία μας δείχνει την ανάγκη η Κομισιόν να θέσει ξεκάθαρου κανόνες για το πεδίο εφαρμογή και τη συχνότητα αυτών των επαληθεύσεων, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και των προγραμμάτων για το πώς υλοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι στην πράξη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ όσοι διαμαρτύρονται για τους υπερβολικά πολλούς ελέγχους, τους συνιστώ να διαβάσουν την σελίδα 49 που λέει ότι ελέγχονται το ένα κόμμα κάτι όλων των έργων, του συνόλου των έργων. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Κον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο, τον κύριο Μπάλκο και την ομάδα του για την εργασία και για την σημερινή παρουσίαση. Η έκθεση που υποβάλλουν αποτελεί καλή βάση για την αντιμετώπιση των αδυναμιών των ε, ταμείων για, τον επόμενο, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η έκθεση σημειώνει κατ' επανάληψη ότι σε ό,τι αφορά την κανονιστική υπερεπιβάρυνση έχουμε πάρα πολύ περιθώριο βελτιώσεων. Εγώ θεωρώ πάντως ότι ε, η υπόθεση αυτή είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η πολιτική στήριξη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράδειγμα από τη Γαλλία με 16 σελίδες ε, το νομοθέτημα, ενώ στη Γερμανία το ίδιο νομοθέτημα είναι 59 σελίδων και στην Πολωνία 28, διορτάται κανεί αν τα πράγματα αυτά είναι αναγκαία. Δείχνει όμως ότι συχνά αυξάνεται η γραφειοκρατία και οδηγεί βέβαια σε αποστροφή εν τέλει και απογοήτευση των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι τελικώς καταλήγουν να προτιμήσουν να παρετηθούν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το οποίο δεν θέλουμε όμως τα μηνύματα που λαμβάνουμε τα ακούμε. Πρόσφατα συναντήθηκα στην περιφέρειά μου, Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, με την Πρωθυπουργό του Κρατηδίου για να δούμε τρόπους να βελτιωθεί η κατάσταση. Ένας τρόπος είναι οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις να διατυπώνονται με απλούστερο και ευκρινέστερο τρόπο, ώστε να υπάρχουν και λιγότερες ερμηνείες που να μπορούν να κάνουν οι χώρες μέλη και επομένως να οδηγούμαστε και τελικώς σε λιγότερη γραφειοκρατία. Η Πρόεδρος μίλησε μόλις για τους ελέγχους. Βεβαίως και αυτό είναι ένα τομέας που πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι δικαιούχοι να μην δέχονται διαρκώς επισκέψεις των ελεγκτών είτε από την ευρωπαϊκή πλευρά είτε από την εθνική διότι βεβαίως εκεί παίζουν ρόλο και αυτά τα πράγματα και αυτό οδηγεί πάλι σε μια αίσθηση ματέωσης και σε μια αίσθηση αποστροφής. Ε, βεβαίως από την άλλη μεριά λέμε ότι καλή εμπιστοσύνη καλύτερο ο Χρειάζεται να εξισορροπηθούν οι ανάγκες αυτές και να εξετάζεται πού πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, ε, αν πρέπει να γίνεται από διάφορα επίπεδα, να είναι πιο ε, ισορροπημένη έλεγχη. Ε, ο κανονισμός Omnibus κάνει και τη διάκριση across reliance κλπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης υποβάλλει καλές προτάσεις στον γενικό κανονισμό. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ θα λάβει υπόψη τι συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά έχω και μια ερώτηση προ το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο. Ποια εντύπωση έχει για τον νέο γενικό κανονισμό και πού θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρξουν βελτιώσει. Σα ευχαριστώ. Ο κ. Νοβακόφ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κον αλλά και τον κύριο Μπάλκο βεβαίως του ελεγκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να τονίσω κάτι, δηλαδή το χρονικό σημείο όπου λαμβάνουμε την ενημέρωση αυτή. Διότι εργαζόμαστε ας πούμε τον τελευταίο μήνα για το CPR και ένα από τα κεφάλαια είναι η απλοποίηση. Εγώ πρέπει να πω χωρίς κανένα δισταγμό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασφαλώς κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός στην πρότασή της και ιδίως όσον αφορά την απλούστευση. Flat rates, ε, απλουστευμένες επιλογές κόστους αποτελούν μέρος της λύσεως και πιστεύω ότι η πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση που βλέπουμε καμιά φορά είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι δικαιούχοι προτιμούν ακόμη να πάνε στην τράπεζα και να πάρουν ένα δάνειο το οποίο θα ξεπληρώσουν με τους τόκους αντί να μπλέξουν με την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και ιδίω όσον αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή τις λεγόμενες νεοφύης, startups. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπάθειες που γίνονται για να επέλθουν αλλαγές, όχι επαναστατικές αλλαγές, αλλά αλλαγές για την περίοδο μετά το 2020. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομάδα υψηλού επίπεδου για την ε, απλοποίηση. Θα έχουμε τα συμπεράσματα και θα μπορέσουν να αρχίσουν να εφαρμόζονται ίσως και του χρόνου, ένα χρόνο πριν από τη λήξη της προγραμματικής περίοδου. Δεν μπορούμε όμως να επιτρέψουμε άλλες καθυστερήσεις. Πιστεύω ότι η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής μπορεί να αναβαθμιστεί και είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα ζητήσει την ενίσχυσή της. Και ιδίω ό,τι αφορά την απλούστευση, διότι η απλούστευση είναι βέβαια περίπλοκη διαδικασία και προσφέρει και τροφή στον ευρωσκεπτικισμό που τα φορτώνουν όλα στις Βρυξέλλες ότι αυτοί ζουν μέσα σε μια φούσκα, δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στο πραγματικό κόσμο κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλογραμμένο το έγγραφο και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για το μέλλον, για την σύνταξη του Γενικού Κανονισμού και τις άλλες διατάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση και ευχαριστούμε και τον κύριο Κον για τις παρατηρήσεις του σε σχέση με αυτό το ενημερωτικό έγγραφο το οποίο θα λάβουμε υπόψη μας. Θέλουμε πάρα πολύ θετική την αναγνώριση των επιτευγμάτων για να θωρακιστούν αυτοί οι εσωτερικοί έλεγχοι, να μειωθεί το ποστό σφάλματος σε σχέση με τα ήδη έχουμε καταφέρει για την πολιτική συνοχή. Και συμφωνούμε 100% ότι η απλούστευση θα πρέπει να θεωρηθεί ως το μέσο για να έχουμε καλύτερη λογοδοσία αλλά και απόδοση. Τόσο αφορά αυτούς τους πέντε τομείς που τονίζει το ελληνικό συνέδριο στο ενήμερο δικό του και τα πέντε αυτά σημεία αφορούν την απλούστευση, την πρότασή μας της 29ης Μαΐου για τη δεσμέτρων της συνοχής. Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία για την απλούστευση στο website της DigiRegio και αναφέρονται εκεί αυτά τα μέτρα πρόταση τη πολιτική συνοχή. Και από εκεί μπορεί να καταλάβει κανεί ότι είναι κάτι το ευρύτερο τελικά η απλούστευση, κάτι ευρύτερο από αυτούς τους πέντε τομεί. Ο στόχος μας ήταν οι δικαιούχη. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο θεωρήσαμε ότι έρχονται κάποιοι κανόνες για τη διαχείριση και για τις αρχές. Νομίζω αυτά είναι αναπόσπαστα δεμένα μεταξύ τους τώρα όσον αφορά τις καθεντήρες γραμμές. Είναι 5% συντομότερο ο CPR από ότι ο 14-20. Κάτι λέει αυτό δεν είναι μόνο ποσοτικό. Επίσης, η αυτογενής νομοθεσία επίσης έχει μειωθεί. Το τα Όλοι οι κανόνες χρειάζονται για τον προγραμματισμό και όλα αυτά προβλέπονται και καλύπτονται εκεί. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Να γίνουν όλα πιο απλά. Έχουμε κάποιες ε, ρυθμίσεις για την απλούστευση των προγραμμάτων όσον αφορά τις εκθέσεις τις σχετικές με τον προγραμματισμό και αυτό αφορά την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, οπότε πρόκειται για θέμα επιλογής τελικά των κρατών μελών ή μπορεί να γίνουν και διαπραγματεύσει. Οπότε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπάρχει κίνητρα τόσο ώστε να υπάρχει τέτοιου είδους εκτονική των προγραμμάτων που να καλύπτονται από το stream, από streamline αντιμετώπιση. Αποσταθμένη δηλαδή. Τώρα, Για όλα θέλουμε να υπάρχουν όμως απλουστευμένοι, ε, κανόνες. Αυτό αφορά και ε, την, την, τον πολλαπλασιασμό των νομοθετημάτων, τον gold plating και τα κρατη βέβαια τελικά έχουν την τελευταία λέξη. Τώρα όσον αφορά κόστος, δαπάνες, η σημερινή ε, ισχύουσα νομοθεσία. Πρόκειται να εξελιχθεί εν ώψη του προγραμματισμού του 2020. πριν για τα flat rate. Πρότεινε τη ευρία χρήση αυτών όπως ε, ανέφερε ο κύριος Νόβακοφ. και τη χρηματοδότηση σε σχέση με τις δαπάνες και εδώ έχουμε φιλοδοξίες για τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Τώρα για τους πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Έχουμε τρεις σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Την απλούστευση των ε, επαληθεύσεων διαχείρισης ακριβώς όπως ε, προβλέπει ο κανονισμός CPR. Αναλογική ρύθμιση για τους ελέγχους σε προγράμματα που έχουν ε, καλή προϊστορία σε σχέση με τους κινδύνους. Επομένως και εδώ έχουμε μείζωνα απλούστευση. Και όσον αφορά διαχείριση και έλεγχο, σας τονίζουμε τον, τους λογιστικούς έλεγχους που μπορεί να έχει η αρχή διαχείρισης και εδώ επίσης μπορούμε να έχουμε περιθωρία πλούστευσης σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Πρόεδρος, συμπάθεια θα πρέπει να προχωρήσουμε και έχουμε και ένα άλλο σημείο σε διάταξη Άρα ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να ξεκαθαρίσετε διμερώς. Θα, θα καλωσορίσω μάλλον τα μέλη της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών για το έγγραφο του ε, Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Γκρέγκο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για το λόγο κύριε Σιγητά, μέλη του Κοινοβουλίου και κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα ενημερωτικό έγγραφο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την πρόταση της ε, Κομισιόν για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πιθανότητα που μου δίνεται, δυνατότητα που μου δίνεται να παρουσιάσω το έγγραφό μας, αφού εγκρίθηκε από το Σώμα. Και αφού δημοσιεύτηκε χθε από το ελεκτικό συνέδριο η σημερινή μου παρουσίαση, θα συμπεριλάβει τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα επικεντρωθώ στη σύγκριση μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων, η πρώτη από το 2014 μέχρι το 2020 και την προτινόμενη από το 2021 στο 2027. Και στο δεύτερο τμήμα θα αναφέρω τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ε, εκπόνηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και στο τελευταίο τμήμα θα προβώ σε ένα follow-up ε, σε σχέση με το πρώτο έγγραφο που είχαμε αρχικά εκδώσει. Λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια να σας παρουσιάσω μία επισκόπηση των πολυάριθμων δραστηριοτήτων του ελεκτικού συνεδρίου σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη σχετική πρόταση. Αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε δύο οριζόντια ενημερωτικά εγγραφά για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Παρουσίασα ένα το Φεβρουάριο και σήμερα παρουσιάζω το δεύτερο που ακολουθεί τις πρότασεις της Κομισιόν. Επίσης, δημοσιεύσαμε μία σειρά εγγράφων τομεακών το που παρουσιάζεται σήμερα και μετά από το δικό μου έγγραφο θα έχουμε άλλη μια σειρά προϊόντων του ελεκτικού συνεδρίου. Όμως αυτή τη φορά θα προετοιμάσουμε τις γνωμοδοτήσεις μας. Ορισμένες εξ αυτών είναι μέρος της νομοθετικής διαδικασίας όταν ε, μας διαβουλεύονται ως μέρος της ε, διαδικασίας. Αυτό αφορά κυρίως τους ίδιους πόρους, την απόφαση για τους ίδιους πόρους και το κράτος δικαίου, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προετοιμάζουμε γνωμοδοτήσεις που μας έχουν ζητηθεί, κυρίως από το Κοινοβούλιο. Αυτό θα συμπεριλάβει τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων για τα τρία ταμεία, το Ταμείο Θαλασσασκελίας το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το Μέσο Διαχείρισης των Συνόρων και Θεωρήσεων και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Κάποιες άλλες γνωμοδοτήσεις ε, ίσως να ακολουθήσουν και για το Ταμείο U-Invest. Μέχρι τώρα δεν μας έχει ζητηθεί όμως. Αυτή, σε αυτή το έγγραφο, το ενημερωτικό, επικεντρωθήκαμε στον προτινόμενο κανονισμό για ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τη σχετική ανακοίνωση, την ε, ανασκόπηση δαπανών και έχουμε αναλύσει και την ίδια την πρόταση, καθώς και τη διαδικασία για την εκπονήση. Το έγγραφο δεν αποτελεί αποτελεσμα ελέγχου, αλλά αποτέλεσμα της ε, επισκόπησης των διαθέσιμων εγγράφων. Στη διαφάνεια αυτή Θέλω να σας υπενθυμίσω ποιες είναι οι κύριες αρχές της Κομισιόν για την ε, προετοιμασία ε, του εγγράφου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, προσθεμένη αξία, απλούστευση, λογοδοσία ε, και ευελιξία. Εδώ στο πρώτο μας έγγραφο εξετάσαμε τις αρχές αυτές σε, όλες, σε όλα τα στάδια του δημοσιονομικού κύκλου, δηλαδή όταν τίθενται οι προτεραιότητες, όταν, όταν εκπονούνται, κατανέμονται οι πόροι ε, και ε, όταν εφαρμόζονται τα προγράμματα και κατόπιν κατά τη διάρκεια των αποτελεσμάτων. Τώρα να πάω στο πρώτο μέρος της παρουσίασης. Στόχος του είναι να συγκρίνει το παλιό και το νέο πλαίσιο. Η πρόταση της Κομισιόν ΕΖΗ αυξήσει για τι προτεραιότητε στην ΕΛΕΑ, την ασφάλεια, τα σύνορα και τη μετανάστευση. Από τη δική μα σκοπιά, αναρωτηθήκαμε αν αυτό προβλέπει μια σαφή σύγκριση μεταξύ των σημερινών και του νέου πλασίου. Και πιστέψαμε ότι χρειάζεται να παρουσιάσουμε αυτή τη συνολική σύγκριση για να έχουμε μια καλή κατανόηση. Γι' αυτό και βλέπετε και το μέγεθος του εγγράφου και ελπίζω το έγγραφο να σας διαφωτίσει για τις προτάσεις της Κομισιόν. Στην επόμενη διαφάνεια, εδώ βλέπετε πώς προσεγγίσαμε το θέμα της συγκρισιμότητας μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων. Δεν είναι κάτι απλό. Υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα. το χάρη, έχουμε τον πληθωρισμό ε, την αξία των χρημάτων στη συγκεκριμένη περίοδο. Στη σημερινή περίοδο 14-20 παρουσιάστηκε σε τιμές του 2011. Έτσι λοιπόν, ε, για να προσαρμοστούμε στις ε, τιμές του 2018, προσθέσαμε πάνω κάτω 19 δισεκατομμύρια. Βέβαια, πρέπει να εργαστούμε και λαμβάνοντα υπόψη τον Brexit. Δυστυχώ, εξακολουθεί να είναι επιτάπητο. Έπρεπε λοιπόν να αφαιρέσουμε περίπου 53 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι το ποσό που εκτιμά η Κομισιόν ότι θα δοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στους δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλη την περίοδο 2014-2020. Η επόμενη προσαρμογή σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Στην τελευταία περίοδο είχαμε ε, περίπου 28 δισεκατομμύρια. Αυτό πρέπει να προσθεθεί για λόγους ε, σύγκρισης και υπάρχει και μια αλλαγή της δομής ε, των τομέων. Αυτό δεν είναι σημαντικό για το συνολικό ποσό, αλλά είναι σημαντικό όταν συγκρίνουμε με μονομένους τομείς του προπολογισμού και προτεραιότητες. Στην επόμενη διαφάνεια προσπαθήσαμε να τονίσουμε τις αλλαγές στις προτεραιότητες ε, δαπανών. Ένας ε, τομέας απλώς άλλαξε όνομα σε πόρους φύση και το περιβάλλον δημιουργήθηκαν όμως νέοι τομεί μετανάστευση, διαχείριση των συνόρων, άμυνα και ασφάλεια και με τα βέλη και τα ποσά. Προσπαθήσαμε να δείξουμε την ε, αλλαγή των προγραμμάτων μεταξύ των τομέων. Μόνο δύο τομείς ε, δεν επλήγησαν, η γεωργία και η διοίκηση. Οι μεγαλύτερες δαπάνες ε, είναι υπό την κοινή διαχείριση. Η κεντρική πρόταση του πλαισίου δεν περιγράφει λεπτομερώ τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θα εφαρμοστούν για την ε, προκατανομή των δαπανών. Παρ' όλα αυτά, κάποιες λεπτομέρειες υπάρχουν στην τομέακη νομοθεσία για τα ταμεία συνοχής και για τη γεωργία. Στην επόμενη διαφάνεια προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε το συνολικό όγκο της πρότασης της Κομισιόν σε τρέχουσες τιμές, τη σημερινή περίοδο αποτελεί 1,387 εκατομμύριο 87 δισεκατομμύρια, ενώ η νέα περίοδος φτάνει στο 1 εκατομμύριο 279 δισεκατομμύρια, αυτό είναι σε τρέχουσες τιμές και αφού εφαρμόσαμε όλες τις προσαρμογές που σας παρουσίασα, Έχουμε πραγματική αύξηση 5% με απόλυτους όρους, ε, συν 53 δις ε, λοιπόν, μεταξύ των δύο προγραμματικών ε, περίοδων και σε σχετικούς όρους για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα έχουμε μείωση από το 1,16 στο 1,11 για την Ευρώπη των 27. Στην επόμενη διαφάνεια θέλω να επικεντρωθώ στη δομή των τομέων του προπολογισμού υπάρχει μείωση στους φυσικούς πόρους και στο περιβάλλον. Έχει ασύμμετρα αποτελέσματα εντός του τομέα. Άμεσες πληρωμές θα μειωθούν κατά 11%, η ανάπτυξη της υπαίθρου κατά 28%, αλλά εδώ πρέπει να είμαι δίκαιος. Συνδέεται αυτό και με το θέμα της ε, πρότασης χρηματοδότηση. Αλλάζει σε χρηματοδότηση στον στην τομεακή νομοθεσία. Επομένως, η επίπτωση στο συνολικό των προγραμμάτων δεν είναι 20% αλλά χαμηλότερο. Και τέλος, ε, για το περιβάλλον και το κλίμα προτείνεται αύξηση κατά 50%. Στον άλλο σημαντικό τομέα, συνοχή και αξίες, ε, τα ταμεία συνοχής ε, αφορούν το Ταμείο Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προτίζεται μία μείωση του 10% και πάλι εδώ έχουμε ασύμετρη προσέγγιση. Για το ΕΤΠΑ υπάρχει προτιμούμενη μείωση 2% για το Ταμείο Συνοχή 45% και για το Κοινωνικό Ταμείο μείωση 7% και το Erasmus ε, Plus συν 92%. Ο τομέας ε, δημόσια διοίκηση θα αυξηθεί κατά 7% από το οποίο το 3% πάει στην ε, διοίκηση των θεσμικών οργάνων ε, και 100% ε, για τα σχολεία και στις συντάξεις. Ο συνολικός αριθμός των νέων είναι 150 δις και το 63 θεωρώ ότι αποτελεί νέε προτεραιότητε εντό υφιστάμενων πολιτικών και το 52 δι είναι προσθέτη χρηματοδότηση. Δηλαδή, για κάθε ευρώ ε, εσωτερική ε, νέα ιεράρχηση ε, έχει βάλει 80 σέντσι κομισιόν για τους νέους πόρους. Θέλω να επικεντρωθώ στην προετοιμασία της πρότασης. Η Κομισιόν προετοίμασε την ε, πρόταση ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, μία εύρωστη διαδικασία. Είχαμε και κάποιες ε, επισκοπήσεις ε, των δαπανών για τις δαπάνες και αυτό εξηγεί τις καθυστερήσεις. Όπως σας είπα, οι επισκοπήσεις για τις δαπάνες συνόδευσε την πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην επόμενη διαφάνεια Προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την θέσπιση των προτεραιοτήτων. Υπάρχει μια τυχή συγκυρία που είναι πέραν του ελέγχου της Κομισιόν. Το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μην ε, έχουμε στρατηγική για το 2030. Η Κομισιόν όμως παρόλα αυτά πρέπει να παρουσιάσει την πρόταση και φυσικά έχει προτείνει το σχέδιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου σε διαβούλευση με του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων το Φεβρουάριο. Για το μέλλον αυτό αποτελεί πρόκληση, γιατί κάποια μέρα θα έχουμε ένα νέο σύνολο προτεραιοτήτων και μέχρι το 2030 πρέπει να ρωτήσουμε αν αυτόν θα συνάδει με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ή πώς θα αντικατοπιστρουν όλα αυτά. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε αναφέρει τις προσδοκίες μας ε, βάσει του σχεδίου προβληματισμού. Ε, βλέπετε εδώ ένα φανάρι, ένα φωτεινό σηματοδότη για να αντικατοπτρίσουμε την ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία και αυτό θα αντικατοπτρίζεται στην ε, ένταση της χρηματοδότησης. Δεν μπορέσαμε να βρούμε το σύνδεσμο μεταξύ της επισκόπησης δεπανών και της πρότασης ό,τι αφορά την προσθεμένη αξία, πιθανότατα η Κομισιόν το έχει πράξει αυτό, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν διαθέσιμα σε εμά. Στην επόμενη διαφάνεια προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις μας. Ε, υπάρχει ένα στοιχείο για ευελιξία. Νομίζω ότι αντικατορίστηκε πλήρως ε, στην πρόταση και υπάρχει και ένα στοιχείο επί του οποίου ε, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος και αυτό αφορά τη γενική προσέγγιση για τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για όλα τα θεσμικά όργανα είτε εντός είτε εκτός ε, της ε, νομικής τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να τελειώσω με ένα, τελευταία διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε τις προκλήσεις και φυσικά έχουν αναπτυχθεί βάσει των προτάσεων του προηγούμενου ενημερωτικού εγγράφου. Να κλείσω λέγοντας ότι στο δεύτερο εξάμεινο του έτους θα παρουσιάσουμε μία σειρά γνωμοδοτήσεων ε, του ελεγκτικού συνεδρίου για την προτεμμένη νομοθεσία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η συγκεκριτής είναι ο κύριος Σάρβαμα. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ιδιαίτερες ευχαριστίες στο ελεγκτικό συνέδριο και το μέλος του κύριο Γκρέγκορ, όλος ιδιαίτερος. Πρώτα θα ήθελα βέβαια να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου για το έργο του ECA συνολικά. Πρόκειται για σε βάθος, ε, σε εξέταση της ε, προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι που με ικανοποιεί ιδιαίτερο είναι ότι το έγγραφο που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ σαφές και ευανάγνωστο. Έχει και επικοδομητικό χαρακτήρα, διότι αναφέρει τις βασικές, τα βασικά ε, ισχυρά σημεία ας πούμε, και τα ασθενή σημεία. Το ελεγκτικό συνέδριο επισημαίνει τις ίδιες αδυναμίες, τις οποίες έχουμε επισημάνει και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον προπολογισμό και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών... δηλαδή και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα, όπως η δική μας ανάλυση. Και ενώ το ελεγκτικό συνέδριο επισημαίνει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι αδυναμίες είναι ανάγλυφες. Ωστόσο, έχουμε μία πρόταση εμείς, προβλέπει περισσότερη ευκαμψία, συμφωνεί ναι, και κάποια απλούστευση, ναι και εδώ, αλλά δεν είναι όμως αρκετά φιλόδοξο θα έλεγα εγώ εν ώψη βέβαια των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμφωνήσουμε με την άποψη του ECA ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προσφέρει ε, ε, πλήρη επισκόπηση των αλλαγών στις δαπάνες. Και εμείς ε, κοπιάσαμε πολύ με την ανάλυση των αριθμών εδώ και καταλήξαμε σε διαφορετικά ποσά. Αυτό εξαρτάται βεβαίως από τις προβλεπόμενες επιπτώσεις του πληθωρισμού, του Brexit κλπ είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Παρόλο που δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις που ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έργο δεν είναι εύκολο να ε, παρακολουθήσει κανείς τους στόχους του, της προτάσεως. Αναμέναμε πρόταση η οποία θα κάλυπτε το κενό της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ελπίζαμε να έχουμε και ενωσιακό προπολογισμό που θα μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους και καθήκοντα που σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών, παρόλο που έχουμε πρόσθετες δαπάνες σε νέους ε, τομείς προτεραιότητας, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι περικοπές ωστόσο είναι δραματικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει πιο φιλόδοξο ενωσιακό προπολογισμό με πιο φιλόδοξους ιδίους πόρους. Όταν τώρα συγκρίνουμε το συνολικό όγκο του τρέχοντος ΠΔΠ με το προτινόμενο, μπορεί να βλέπουμε μεγαλύτερα νούμερα, δεν βλέπουμε όμως ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και παρόλη την αύξηση των δαπανών, μειώνεται η συνεισφορά στην βάση του ΑΕΠ. Σημειώνει επίσης το ελεγκτικό συνέδριο ότι ίσως έχει χρησιμοποιήσει κάποια νούμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς της. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει, κάνει να φαίνονται οι περικοπές μικρότερες και οι αυξήσει περισσότερες, μεγαλύτερες. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές περικοπές και οι νέες προτεραιότητες δεν κερδίζουν τόσο πολύ σε αύξηση δαπανών. Πέραν αυτού, όπως τονίζει πάλι το ελεγκτικό συνέδριο, η πρόταση για το ΠΔΠ χρειάζεται περισσότερη έμφαση στην ε, ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Έχουμε φιλοδοξίες, όμως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στερείται συγκεκριμένων δικτών για την ε, προσθέμενη αξία των δαπανών. Εδώ θέλω να τονίσω την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και ιδίω το αίτημα για, για σημαντικό εξυγχρονισμό και επανασχεδιασμό του προϋπολογισμού στη βάση ε, μετρήσεων της επίδοσης, κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί υπόψη. Αναφέρονται και οι προκλήσεις, τις οποίες εγώ εκλαμβάνω ως συστάσεις. Και νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσε να είχε φανεί και λίγο πιο τολμηρό και να είχε καταστήσει τις συστάσεις αυτές σαφέστερες και να τις καταστήσει σαφείς ως συστάσεις το ελεγκτικό συνέδριο. Τέλος, η ειλικρινή συγχαρητήρια στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό το έγγραφο που έχει υποβάλει δεν είναι μεν τέλειο, είναι όμως πραγματικά κατανοητό και κάτι που μπορεί πραγματικά να συσταθεί η ανάγνωσή του από όλους όσοι λαμβάνουν αποφάσεις και όχι μόνο, αλλά και από τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο, ενεργότερα στην διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ και πάλι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ιδίω το μέλος του κ. Γκρέγκορ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, σας παρακαλώ να είστε σύντομε και σύντομοι, δεν έχουμε πια πολύ χρόνο. Είναι Θέλω να ευχαριστήσω απλώς το Ελληνικό Συνέδριο, διότι άμεσα αντέδρασε και μας ε, γνωμοδότησε. Πρόκειται για την πρώτη μας συζήτηση εδώ. Μπράβο για την ε, ταχύτητα. Είμαστε σε πρώτη ανάγνωση. Μήπως μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξής. Και εγώ προβληματίζομαι. Λέμε για έναν προϋπολογισμό συνδεδεμένο με την αποτελεσματικότητα. Θέλουμε εις βάθος να δούμε τι γίνεται, πώς θα μπορούμε να έχουμε κάποιες ενδείξεις, κριτήρια για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει καλύτερα τι γίνεται. Και έχουμε και για το επόμενο ΠΔΠ τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να δούμε τι στρατηγική θα χαράξουμε για τα επόμενα χρόνια. Είναι δύσκολο, είναι ρηψοκίνδυνο μετά τη χρηματοοικονομική κρίση να έχουμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα μέσω ή μάκρο πρόθεσμου. Γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο της. Αλλά βέβαια θα πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να ασκούμε έλεγχο και να κάνουμε αξιολόγηση για τις επιδόσεις για τα αποτελέσματα. να μας πει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη γνώμη της. Να μας πει για αυτά τα κριτήρια. Αλλά μας πει και το ελληνικό συνέδριο τι πιστεύει, τι γίνεται με την νομοθεσία που θα εφαρμοστεί σχετικά. για τους σχετικούς κανονισμούς. Γιατί εμείς ε, νομοθετούμε από τη μία, αλλά από την άλλη τα πράγματα γίνονται λένε και πιο δύσκολα. Merci, Madame la Présidente. Je remercie aussi, euh, Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και το Εθνικό Συνέδριο για τα όσα μας ε, είπε. Αν μπορεί κάποια στιγμή τώρα κοντά να μας ε, πει τη γνώμη του Εθνικού Συνέδριου για την μεθοδολογία. Δεν, ναι, δεν μιλούμε τώρα για τα ποσά. Να σας εξηγήσω ότι ενώ έχει μια μεθοδολογία Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την ονομάζουμε top-down από την κορυφή προς τη βάση ε, αφαιρετική ας την πούμε. Δίνει 1% για τις ε, πληρωμές, αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη και κατόπιν γίνεται η κατανομή για τις προτεραιότητες. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Και αυτό έχει πίεση να γίνει το Συμβούλιο. Ωραία. Να όμως τι θέλουμε για ε, την ερωτική πολιτική. Τι θέλουμε για την πολιτική συνοχή. Πόσα χρειαζόμαστε για την άμυνα. Πόσα χρήματα για το Erasmus Plus, για την ε, νεολαία. Κάνουμε το άθροισμα και βλέπουμε μόνο τι προκύπτει. Να, μια καλή μεθοδολογία. Όμως τι πρεσβεύει το ελληνικό συνέδριο για αυτά τα ποσά, για αυτή τη μεθοδολογία. Άλλο, διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πολιτική συνοχή με τις περικοπές της κλπ. Αλλά με κάποιες σταθερές τιμές από την άλλη. Όμως τελικά έχουμε περικοπές και υψημένες δαπάνε και για την ε, και για τη Γεωργία. Και άλλα ήθελαν τα κρατη υιοθέτησε αυτή τη μεθοδολογία των σταθερών τιμών. Να, επομένως πώς προέγυψε μία σύγχυση. Τι είναι τελικά, οι τρέχουσε τιμέ ή σταθερέ τιμέ που θα χρησιμοποιήσουμε. Προσθέμενη αξία. Πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι ορίζεται προσθέμενη αξία, κάτι για το οποίο μιλάει όλο ο κόσμο. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει έναν ε, ορισμό. Μπορεί να μας βοηθήσει, να μας πει τι πάει να πει ε, προς αξία. Εύκολο να λέμε ότι θέλουμε όλα τα προγράμματα να δίνουν προσθέμενη αξία. Τελευταία, ευελιξία. Ναι, αλλά μέχρι ποιο σημείο. Το μάξιμο ευελιξία σημαίνει να έχουμε μόνο μία κατηγορία, μόνο ένα κεφάλαιο, μόνο ένα κονδύλι στον προπολογισμό. Να, η μεγίστη ευελιξία. Άρα ναι στην ευελιξία, αλλά χρειάζεται σαφήνεια, χρειάζεται διαφάνεια για το πώς λειτουργεί. Στρατηγική, ναι, 2020 συν, οι στόχοι παραμένουν, αλλά έχουμε νέες προτεραιότητες, άμυνα, μετανάστευση, ασφάλεια. Στα αγγλικά θα συνεχίσουμε, λέει η πρόεδρος, το 12.30 σταματά η δερμηνία. First of all, I would like also to thank for the comprehensive report which has been made for this presentation. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή. Αν δούμε τις λεπτομέρειες, βλέπουμε το τμήμα που αφορά τις δαπάνες αλλά και τα έσοδα για το επόμενο πολιτές πλαίσιο αλλά και ε, τη συγκρισιμότητα με τις σημερινές παραμέτρους. Τα γραφήματα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να καταλάβουμε τις αλλαγές ε, και το σκοπό των συλλογών στη χρηματοδότηση σε διάφορους τομείς ε, για τον επόμενο προγραμματική περίοδο. Βάσει των στοιχείων που μας παρουσιάστηκαν και που μας εστάλησαν, Νομίζω ότι χρειάζονται ορισμένε διευκρινήσεις. Το πρώτο είναι η ανάγκη για μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμπεριλαμβάνει όλες ε, τις ε, ε, ε κονδυλία σε προτεραιότητες και τη θέσπιση στρατηγικών στόχων. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί σε μια μεγαλύτερη περίοδο. Παραδείγματο χάρη, αναφέρομαι στη στρατηγική για το 2030 που θα μπορούσε να είναι κινητήριο δύναμη για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Εξακολουθούμε να μην έχουμε μια στρατηγική για την επόμενη δεκαετία. Μιλάμε για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εξακολουθούμε όμως να μην έχουμε μια τέτοια στρατηγική και νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό να έχουμε μια τέτοια στρατηγική και να μιλάμε για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εδώ θα σταματήσει η διερμηνία. Σας ευχαριστούμε. The second concerns establishing public audit mandates for all EU-related bodies, having regard the lack of opportunity for audit of some EU bodies, as well as the bodies established through agreements outside the, outside the EU legal order.